Uh, Γεια σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη που σας ε, καθυστέρησα. Μόλις ε, ε, κατέφθασα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε μια διάσκεψη με τον Αντιπρόεδρο Ψεύσκοβιτς για τα ενεργειακά και την περιφερειακή συνεργασία και όλα τα συμπαραμαρτούντα ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ας προχωρήσουμε στην ημερησία διάταξη της Επιτροπής μας, έγκριση αυτής. Έχετε τίποτα σχόλια? Όχι, κανένα. Ωραία. Ούτε ειδικέ ανακοινώσει έχω να σα κάνω εγώ. Η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 10η και 24η Σεπτεμβρίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσει μέχρι το τέλος συνεδρίας θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Α περάσουμε αμέσω στο 4. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδει παραμέτρους. Η συγγητής μας είναι ο κ. Μίχο Μπόνι. Και σκιώδης αναφέρονται εδώ στον κατάλογό μου. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτή την πρόταση αναθεωρημένου κανονισμού για την επισήμανση των ελαστικών ε, το Μάιο του 2018 σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμων. Θα παρακαλέσω τον εισηγητή να πάρει το λόγο για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ε, κύριος Μπόνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και επίσης ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσής μου. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα αναθεώρηση της συνολικών επιδόσεων και της ποιότητας των ελαστικών που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντική η συνεισφορά αυτή και για την οδική ασφάλεια, γενικότερα την ασφάλεια των μεταφορών, αλλά και την κατανάλωση καυσίμων ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι έχει σημασία αυτό απόλυτη, το αυριανό σύστημα μεταφορών να είναι καθαρό, αποτελεσματικό και ασφαλές για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό όλοι αυτοί οι υψηλοί στόχοι απαιτούν την πλήρη προσήλωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενδιαφερομένων και συμφεροντούχων και σε ό,τι αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Η πρόταση ε, επιτρέπει ε, να αναγράφει στην επισήμανση ε, κάποιες προφορίες για τα λάστιχα χιονιού και τα χειμερινά λάστιχα. Πολλέ φορέ δεν τα βλέπουν καν οι ε, καταναλωτές τα λάστιχα που πρέπει να αγοράσουν γιατί είναι κάπου αποθηκευμένα και ε, θα παραγγέλνουν από το διαδίκτυο. Κανονικά θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές ε, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο προμηθεύονται τα ελαστικά του οχήματος. Επίσης, θα ενταχθούν και τα ελαστικά στην βάση δεδομένων για την καταγραφή των προϊόντων ε, στο 1369 το 2017 για να βελτιωθεί η ε, παρακολούθηση εποπτεία της αγοράς και ενημέρωση των καταναλωτών. Καλωσορίζω την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερα στοιχεία όπως είναι η ηλικία και η φθορά των ελαστικών. Θα είναι πιο αξιόπιστες οι παράμετροι όμως αν μπορούν να ελέγχονται καλύτερα. Γι' αυτό δεν θα... Ε, επίσης, η, ε, η ετικέτα στο μέλλον ε, και επίσης με καταξιδότηση πράξης θα αναθεωρείται η οδηγία έτσι ώστε να περιλαμβάνεται η χιλιομετρική απόσταση που έχουν διανύσει και η φθορά που έχουν από την τριβή. και το χιλιομετρικό προσδόκιμο του κάθε ελαστικού. Ε, το 30% αφορά σε 5 ε, εκατομμύρια λάστιχα. Επίσης, η αναγόμωση είναι κάτι που επιτρέπει να κάνουμε οικονομίες ενέργειας, ε, εξυπηρετεί την κυκλική οικονομία και μειώνει και το βουνό των αποβλήτων που έχουμε τις ποσότητες αποβλήτων. χρειάζεται πολλή δουλειά για να ενημερώνονται οι καταναλωτές ε, για να συνειδητοποιήσουν τι ελαστικά αγοράζουν, ποια είναι η ποιότητά τους. Ε, τα ελαστικά τα οποία πολλούνται με τα νέα ιοταχή ή με διαφορετικό τρόπο. Χρειάζεται μεγαλύτερη υποπτία στην αγορά και δημιουργία καλύτερων πλατφορμών για να μπορέσουν οι αρχές να συντονίζουν τις δράσεις τους και να υλοποιούν και να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Γι' αυτό η σήμανση ε, των ελαστικών επισώτρων είναι σχετικά νέο μέτρο και εργαλείο και είναι πολύ νωρίς ε, από τώρα για να αλλάξει τελείως ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σήμανση. Να γίνουν κάποιες αλλαγές αλλά να μην ε, ανατραπεί ριζικά το σύστημα. Γι' αυτό προτείνω στις τροπολογίες το μέγεθος της σήμανσης, της ετικέτας δηλαδή, να είναι το ίδιο αλλά να έχουμε επιπλέον πληροφορίες για την ε, πρόσθεση ε, στο πάγο ή στο χιόνι ε, κτλ. The same, but with new, with Το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Για να αλλάξει αυτή χρειάζεται συλλογική προσέγγιση στην Ευρώπη, όπου εθνικοί και ευρωπαϊκοί θεσμοί ή οργανώσει πολιτών, αλλά και αστυνομία και όσοι ασχολούνται με ε, την οδική ασφάλεια να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τα ελαστικά και τις παραμέτρους τους. Και τέλος, ε, προτείνω να παραμείνει η σήμανση ε, σε ό,τι αφορά την αντίσταση των ελαστικών ε, και κάποιες άλλες παραμέτρους, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα χρονοδιάγραμμα πάρα πολύ φιλόδοξο, επειδή έχουμε νέε παραμέτρους, αλλά και μια διαδικασία καταγραφής. Ε, αυτό το συζητήσαμε με διάφορους ενδιαφερομένους επαγγελματίε επαγγελματίες του κλάδου και στη δική μας ε, ομάδα εργασία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχουν προσδοκίες για τη μελέτη αντικτύπου που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες και μας δημιουργούν κάποια ερωτηματικά. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με λογική, με την κοινή λογική, για να φτάσουμε με σταθερότητα στους όχους ε, απαγκίστρωσης από το διοξίδιο του άνθρακα στις μεταφορές, διατηρώντας την ασφάλεια με τις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες, να τους βοηθούμε και να έχουν ε, μια ενημέρωση για να επιλέγουν με τα λόγου γνώσεως τα ελαστικά τους και να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις. Και ο αντισηγητές τώρα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Μαχτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί η εργασία, η έκθεση που μας προτείνει με βρίσκει καταρχάς σύμφωνο. Θα ήθελα να θέσω μερικά σημεία. Η Επιτροπή ε, Βεβαίως συμφωνούμε για να βελτιώσουμε την επισήμανση, τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων, την ε, μείωση κατανάλωση καυσίμων, αλλά και την ε, εκπομπή, ε, ε, τα μικροπλαστικά. Συμφωνώ με την πρόταση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει όμως να προσέξουμε, γιατί μερικές φορές το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Σε ό,τι αφορά την σήμανση, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε ένα ενιαίο τύπο σήμανσης. Ο καταναλωτής είναι συνηθισμένος στις ε, παρούσες ετικέτες, ε, σημάνσεις ε, που είναι πολύ πιο αναγνώσιμες από αυτές που προτείνει η Επιτροπή. Θα πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την πρόσπιση και το χιλιομετρικό προσδόκιμο. Εκεί που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το σημείο που η Επιτροπή κάνει τη διαπίστωση ότι στις κατηγορίες Α και Β δεν θα πρέπει να ε, προσθέσουμε μία κατηγορία όπως έχει γίνει στις οικιακές συσκευές το α συν συν. Απλά και μόνο θα Πρέπει οι κατασκευαστές να βελτιώσουν την ποιότητα αυτών των κατηγοριών. Προσέξτε, προσέξτε για το θέμα των τιμών. Πολύ συχνά η τιμή είναι το πρώτο κριτήριο που καθορίζει την επιλογή του καταναλωτή. Εκεί θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να μην υπάρξει έκρηξη των τιμών. Άλλες ε, τροπολογίες που κατέθεσα φορούν την ίχνηλασιμότητα της ε, προέλευσης ε, των ελαστικών. Πολλοί κατασκευαστές έχουν συνάψει συμφωνίες και θα πρέπει να προσέξουμε να υπάρξει μία βιώσιμη διαχείριση σε ό,τι αφορά τη χρήση χημικών προϊόντων που δεν θα επηρεάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό ισχύει και για την παραγωγή και για τη διάρκεια των ελαστικών. Αυτά θα ήθελα να πω σε γενικές γραμμές. Συμφωνώ με την πρόταση του συγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όταν υπάρχει συμφωνία, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Ο κύριος Νταλούντε, μέρος των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Ε, δύο προβληματισμούς έχουν οι πράσινοι σε ό,τι αφορά την πρόταση της ε, Επιτροπής. Λογότυπος για το χιόνι και τον πάγο που συμπεριλαμβάνεται. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν είναι σωστό. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μία ε, ένα στοιχείο που να αφορά η πρόσφυση. Ένας απλός λογότυπος χωρίς κλίμακα δεν είναι επαρκής γιατί αυτό διακυβεύει την ασφάλεια των πολιτών. Δεύτερον, η πρόταση δεν ε, ε, προωθεί συγκεκριμένους δείκτες όπως χιλιομετρικό προσδόκιμο και πρόσφυση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που παίζουν αυτά τα περιβαλλοντικά σημεία αλλά δεν καθορίζει κάποια προθεσμία. Συνεπώς προτείνουμε να επιταχύνουμε την επεξεργασία εναρμονισμένων κειμένων για το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την πρόσφυση. Περιμένουμε την συζήτηση αυτών των προτάσεων με τους χιώδεις εισηγητές και θα το επιθυμούσαμε να επιτύχουμε μία συμφωνία η οποία προστατεύει και τους καταναλωτές αλλά και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφα για τις παρατηρήσεις σας. Εξ ονόματος της ε, Γκουε, παρακαλώ ρικοχής. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις και από μένα. Καταρχάς η τεχνική πτυχή των όσων συζητάμε. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφής. Ο καταναλωτής θα πρέπει να καταλαβαίνει τι αγοράζει. Δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε πολλά δεδομένα διαφορετικά, δεν θα εξυπηρετείται ο στόχος του. Και μία υποσημείωση. Η πρόσφυση ενός ελαστικού επίσωστρου στο, σε υγρασία, στο χιόνι, στον πάγο, εξαρτάται από το τι υπάρχει από κάτω. Τι είναι άσφαλτος, τσιμέντο, ε, ή αναγωμωμένη άσφαλτο στην οποία έχουν συμπεριληφθεί και κομμάτια από ελαστικά. Αυτή θα είναι μια ελαστική επιφάνεια που προσφέρει μεγαλύτερη πρόσφυση και ε, κατά συνέπεια οι επιδόσεις ε, του ελαστικού θα είναι καλύτερες. Για το λόγο αυτό, προκαταρακτικά συμφώνησα με την έννοια του γραμμικού κώδικα, του barcode, για κάθε ελαστικό έτσι ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να συγκρίνει τα ελαστικά μεταξύ τους και να συγκρίνει και την ποιότητα των ελαστικών, αν είναι για το καλοκαίρι, αν είναι για το χειμώνα ή αν είναι πλέον κατάλληλα για χρήση στη βροχή. Αλλά και ποιο είναι το χιλιομετρικό προσδόκιμο. Και μετά ε, ένα άλλο θέμα είναι το σχέδιο στα ελαστικά και αυτό επηρεάζει το περιβάλλον. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μαρτέν όταν αναφέρεται στη σημασία της πρώτης ύλη και της πηγής των πρώτων υλών. Θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζουν το περιβάλλον. Εγώ θα ήμουν υπέρ μιας απλής ετικέτας που θα μας είπε, θα, που θα μας λέει τι είδους ελαστικό είναι και όλα τα υπόλοιπα υπόλοιπα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό και θα πρέπει σε αυτά να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Όταν μιλάμε για περιπτώσεις που θα πρέπει να υπάρχει η σήμαση και το πώς θα μπορεί να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα στις διαφημίσεις θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται μία εικόνα. Θα μπορούσε κανείς να κλικάρει επάνω και να παίρνει περαιτέρω στοιχεία γιατί ενδεχομένω οι ηλεκτρονικές διαφημίσει μπορεί να είναι ακριβές. Αυτή είναι αυτή λοιπόν η λύση. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές ε, προσδοκίες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τις ικανοποιήσουμε όλες. Εκ μέρου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ο κύριος ε, Λουιλτζή, το συγγνώμη για την προφορά ήταν ενδεχομένως λανθασμένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Περίπου το πετύχατε το όνομά μου. Μη σα απασχολεί. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το λόγο και επιτρέψτε μου να αντιδράσω σε αυτή τη συζήτηση πάνω στο σχέδιο έκθεσης που μόλις ε, παρουσιάστηκε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους ευρωβουλευτές για την στήριξη τους στην πρότασή μας. Γνωρίζω πως ε, θα συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες για το χιόνι, για τον πάγο, για τη σταθερότητα και την ε, διανηθής απόσταση καθώς και την τριβή στα ελαστικά. Και τώρα, ακούστηκε ότι θα έπρεπε η πρόταση αυτή να, είναι, να έχει γίνει νωρίτερα ή αργότερα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και πρέπει να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία για να το κάνουμε πραγματικότητα. Η πρόταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα να ε, μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της πρότασής μας. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε από τον κύριο Μπόνι, τον εισηγητή, είναι η μεγάλη σημασία της βάσης δεδομένων. Πρέπει να είναι προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό. Αυτό αναφέρθηκε και από άλλους ευρωβουλευτές, έτσι ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά και να μπορούν οι καταναλωτές να ενημερώνονται για τις επιδόσεις των ελαστικών που επιλέγουν. Είναι επίσης σημαντικό η βάση αυτή δεδομένων να συμπεριλαμβάνει διάφορα τεχνικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των ε, ελαστικών με τις προδιαγραφές έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Μετά ακούσαμε ε, για, τη, για τους τύπους, για την κατάταξη από τον ε, κύριο Μπόνι και τον κύριο Μαρτάνη. Να πω πως πράγματι η πρότασή μας εμπνεύστηκε από τον ε, γενικότερο κανονισμό για την ε, ενεργειακή σήμανση. Οι ανώτερες τάξεις θα είναι σχεδόν άδειε, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό, χρειάζεται, γι αυτό δεν χρειάζεται ίσως να βιαστούμε τόσο πολύ για την αλλαγή στις ανώτερες κλάσεις η το 90% των ε, τύπων ελαστικών ανήκει στις τρεις ε, ανώτερες τάξεις, οπότε νομίζω πως δεν χρειάζεται κάποια αναδιαμόρφωση των τάξεων αυτών. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα σχόλια για την ε, συμπερίληψη της βιωσιμότητας, ακούστηκαν μερικά παραδείγματα. Βέβαια να πω πως υπάρχουν και ανησυχίες για υπερφόρτωση του συστήματος, για να μην υπάρχουν υπερβολικές πληροφορίες, χρειάζεται να διατηρηθεί κάποια ισορροπία στην επισήμανση. Τέλος. Αυτά είχα να πω νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Μπόνι για κάποια καταληκτικά σχόλια. Α, όχι, θέλετε να τοποθετηθείτε. Παρακαλώ, έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Λάγκεν. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, η έκθεση γενικές γραμμές είναι αρκετά καλή. Πρώτον, να πω πω έχω την πρόθεση να υποβάλω ορισμένε τροπολογίες που αφορούν το γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα άρθρα 4.3 και 6.4 προβλέπει ε, αυστηρότερες προδιαγραφές. 6.2 και 4.3. Ο κύριος Μπόνι έχει κάνει σωστές παρατηρήσεις, μεν όμως η τροπολογία 4 τροποποιεί κάπως ε, τα πράγματα. Αναφέρεται στο διαφημιστικό υλικό. θα πρέπει να αναφέρω ορισμένε πληροφορίε και στο διαφημιστικό υλικό, σε πλακάτα, α πούμε, κτλ. Μετά, η τροπολογία 9. Ο κύριο ε, εισηγητή αναφέρεται στην οπτικοακουστική διαφήμιση, όμως ε, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, για παράδειγμα διαφημίσεις στο διαδίκτυο κτλ. Ε, θα προτιμούσα να διαγραφεί αυτή η τροπολογία, όπως και η τροπολογία 15, όπου συμπληρώνονται κάποιες πληροφορίες, για παράδειγμα, στις επιγραμμικές ε, πληροφορίες ε, που θα πρέπει κάποιος με το ποντίκι του να σκρολάρει προς τα κάτω ή προς τα... Αυτό το θεωρώ περιττό και υπερβολικά ε, λεπτομερές. Γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσω τρεις τροπολογίες σχετικά με αυτά. Τώρα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εμποδίσει ε, την διαφήμιση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, ασχοληθούμε με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία. Όχι μόνο συμπλήρωσαν την παρουσίασή μου, αλλά και με ενέπνευσαν για να συνεχίσω με την αναφορά του στη βιωσιμότητα, για παράδειγμα, ή την χρήση των διάφορων κατηγοριών. Καθώς επίσης και με τα σχόλιά τους για το πώς η πρόταση αυτή θα επηρεάσει τις τιμές. Νομίζω πως μπορούμε να προχωρήσουμε καλά με αυτήν την ε, μορφή συνεργασίας. Ο συνάδελφος επίσης είχε τις προτάσεις του για τη διαφήμιση και τον ευχαριστώ. Νομίζω πως μετά τις ε, τροπολογίες θα ξεκινήσουμε δουλειά, θα τις εξετάσουμε μία-μία για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές, αλλά και να στηρίξουμε την βιομηχανία. χρειάζεται φυσικά να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις απαιτήσει για καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα ελαστικά για χιόνι, για πάγο και για ψύχος. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο 12 το μεσημέρι προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Η εξέτασή τους θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 7 Ιανουαρίου. Επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, σημείο 5 θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας που συμπληρώνει τον μηχανισμό γειτονία ανάπτυξη και συνεργασία σε βάση τη συνθήκη Ευρατόμ. Η εισηγητή είναι ο κύριο Ουρούτσεφ. Η πρόταση, το σχέδιο έκθεση γίνεται στο πλαίσιο του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και συμπληρώνει το που δούμε διάφορε δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στα πλαίσια, στο πλαίσιο της συνθήκης Ευρατών. Κύριε Συγητή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει μια συνέχεια στο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας στη γειτονία της αλλά και σε όλο τον κόσμο. Από την εποχή των ατυχημάτων στο Τσερνόμπιλ και στη Φουκουσίμα οι συνέπειες στην παγκόσμια πολιτική για την πυρηνική ασφάλεια είναι αισθητέ. Χρειάζεται να συμπληρωθεί το, ο ευρύτερος μηχανισμός γειτονίας και διεθνούς συνεργασίας λοιπόν και να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την ε, πληροφόρηση, την παρακολούθηση και την ε, ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η εναρμόνιση των κανόνων είναι ένα σημαντικό βήμα προς την απλούστευση αυτών. Και το Ευρωπαϊκό Μέσο Πυρηνικής Ασφάλειας θα προωθήσει κανόνε κανόνες, πρότυπα και πρακτικέ ε, πυρηνική ασφάλεια και σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τις διατάξει της συνθήκης Ευρατόμ και με τρεις οδηγίες που γνωρίζουμε πολύ καλά για την προστασία από ραδιενέργεια, για την πυρηνική ασφάλεια και για την ασφαλή διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και αναλαιοθέντων καυσίμων. Το σχέδιο έκθεσης τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας και της εφαρμογής αυτής ε, κανόνων για την πυρηνική ασφάλεια, καθώς και προτύπων για αυτή, στην άμεση γειτονία της Ένωσης. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να αντιμετωπίσει πιο ολοκληρωμένα την παρακολούθηση των ε, πυρηνικών καταστάσεων στην άμεση γειτονία της Ένωσης από την ε, πρώτη και όλα στιγμή τα ενδεικτικά πολιτή προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για ε, τις ε, διεξαγωγές ανάλυσης κινδύνου, τις ασφάλειες των εγκαταστάσεων, την εφαρμογή των κανόνων που θα προκύψουν και ε, για τα μέτρα παρακολούθησης. Αυτά τα πολιτή ενδεικτικά προγράμματα θα φορούν χώρες που λαμβάνουν οικονομική στήριξη υπό τον εφιστάμενο κανονισμό, έτσι ώστε εκείνα να μπορέσουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τι συμφωνίε τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, για τη δέσμευση τους ε, στο να τηρούν τις ε, διεθνείς συνθήκες και τα διεθνή πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας καθώς και για την εφαρμογή των ε, σχετικών μέτρων. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε προκαθορισμένους συγκεκριμένους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να βασίζονται σε επιδόσεις, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, έτσι ώστε να αυξηθεί η υπευθυνότητα και η λογοδοσία από τις ε, χώρες αποδέκτες της οικονομικής στήριξης και όχι μόνο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας. Αυτές είναι σε γενικέ γραμμές οι κυριότερες προσθήκες στην πρόταση της Επιτροπής και θα χαρώ πολύ να λάβω τις προτάσεις των συναδέλφων για βελτίωση του σχεδίου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε, opening remarks. για τα εισαγωγικά σα σχόλια. Από του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε. τώρα το λόγο έχει ο κύριο Γκάιο και ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε απολύτω με τον εισηγητή ότι η πυρηνική ασφάλεια στι τρίτε χώρε μετά από τα πυρηνικά ατυχήματα που γνωρίσαμε στο παρελθόν ε, ε, ε, πρέπει να είναι σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η θέσπιση και η τήρηση ε, ε, ψηλότητα των προδιαγραφών θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την προστασία των πολιτών και ε, του περιβάλλοντος. Εγώ δεν είμαι οπαδός της πυρηνικής ενέργειας, αλλά ως καλός δημοκράτης κατανοώ ότι άλλες χώρες έχουν λάβει άλλες αποφάσεις. Ωραία, εν τη αυτή περιπτώση θα πρέπει όμως να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλής αυτή η λειτουργία για να μην απειλούν τους δικούς τους πολίτες και τους πολίτες των γειτονικών χωρών και των περιβάλλων Καλωσορίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μερικά σημεία ε, δεν έχουν ληφθεί επαρκώς ε, υπόψη και καθόλου. Σε αυτό συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με τον εισηγητή και τον ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο έκθεσης. Συμφωνούμε για τα stress test και πόση σημασία έχουν αυτές οι δοκιμές ε, αντοχής και οι διεθνείς συμφωνίες και συνεργασία με διεθνείς θεσμούς όπως είναι ε, η Διεθνής Υπηρεσία ε, Ατομικής Ενέργειας. Ε, το σχέδιο του κανονισμού του Συμβουλίου δεν προβλέπεται στην πρόταση, δεν αναφέρεται, θα πρέπει όμως και οι υψηλέ προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας θα πρέπει να είναι η βάση ίδια της δράσης μας σε τρίτες χώρες και της συνεργασίας. Άλλο στοιχείο που υπήρχε στο προηγούμενο μέσον και τώρα αναφέρεται μόνο σε μια αιτιολογική σκέψη είναι τα ειδικά μέτρα που μπορεί να προωθεί και να ενισχύει αυτό το μέσο. Ε, παρακαλώ και προτείνω να συμπεριληφθεί και στο νέο μέσο το, το παλιό σύστημα και να δούμε ποια μέτρα μπορούν να χρηματοδοτούνται ή να προωθούνται. Και τρίτες χώρες να κληθούν να τα ακολουθήσουν όλα αυτά, αλλά και τιμή διάδοση των πυρηνικών και να δεσμευτούν διεθνώς και να υπογράφουν ε, συμφωνίες και συμβάσεις που υπάρχουν για την πυρηνική ασφάλεια. Δεν σύμφωνο με τους αμυγός ποσοτικούς δείκτες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μέτρηση των ε, επιδόσεων. Θα πρέπει να είναι και ποσοτικές και ποιοτικές. Δηλαδή οι ε, ε, υλοποίηση. Υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που ζητεί η Σύμβαση του Όρους, αρχούς που θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη και προφανώς και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, ο κανονισμός αναφέρεται στο μηχανισμό δανειοδότησης του Euratom, τη διευκόλυνση αυτή. Ε, τι είναι αυτό, αφορά τα 300 εκατομμύρια που προβλέπονται εκεί ή κάτι άλλο. Η κυρία Ριβαζή από την πλευρά των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ώστε λοιπόν έχουμε ένα ενδιαφέρον μέσο ευρωπαϊκό συνεργασία, μηχανισμό με τι τρίτε χώρε για την πυρηνική ασφάλεια. Όμω, ένα από τα πρώτα στοιχεία, γιατί είμαστε και βουλευτέ, είναι ότι παραπέμπεται στη συνθήκη Ευρατόμ. Δηλαδή, θα βοηθήσουμε τρίτες χώρες να βελτιώσουν την πυρηνική τους ασφάλεια, ερήμην τελείω του Κοινοβουλίου. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε τροπολογίες για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συναπόφασης. Έτσι, ε, ώστε όταν επενδύουν στη Ρουμανία, Βουλγαρία, στη Λευκορωσία, στην Ουκρανία, να είμαστε και ενημερωμένοι, αλλά και εκτός από γνωμοδότηση, να παίρνουμε και αποφάσεις ως βουλευτές. Στη συνέχεια έχετε καθέσει κάποια άρθρα για τη σημασία ε, όλων αυτών ε, για τις τρίτες χώρες και αυτά που συμβαίνουν, ο παροπλισμός των πυρηνικών ε, εγκαταστάσεων, η αποκατάσταση των παλιών εγκαταστάσεων που είναι μολυμένες, ας πούμε κάποια παλιά ορυχεία ουρανίου, εμφανίζουν τεράστια ρήπανση και θα πρέπει να αποκατασταθούν γιατί μετά θα υπάρξει πρόβλημα στη γεωργία και ευρύτερα προβλήματα. Αυτό δεν ε, καλύπτεται παρκώς. Υπάρχουν κάποιε πραγματικότητε σήμερα που είναι πάρα πολύ σημαντικέ να υποστηριχθούν τα προβλήματα, να λυθούν τα προβλήματα ρήπανση. Μετά έχουμε τροπολογίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τι μέτρα θα λαμβάνονται σε περίπτωση που δεν γίνονται σεβαστά. Ε, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται, λέτε, σε διαβούλευση και διάλογο με τις τρίτες χώρες. Αλλιώς θα σταματάει η χρηματοδότηση. Κάτι άλλο που είπαν κάποιοι προλαλήσαντες, ε, χρειάζονται και γενικά κριτήρια για να εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες που θέλουν να συνεργάζονται με την Ένωση. Αν επιθυμούν λοιπόν να συνεργάζονται θα πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές αρχές, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, τις αντίστοιχε συμβάσει, τα πρωτόκολλα, ε, συμβάσει άρχους κλπ. Γιατί μην τους δίνουμε λεφτά και μετά δεν έχουμε ε, κριτήρια επιλεξιμότητας. Και τέλος διαφάνεια. Έχει σημασία οι πυρηνικές εγκαταστάσεις να σέβονται τα πρότυπα διαφάνειας και να ενημερώνεται το κοινό όσο και να συμμετέχει στις συζητήσεις. Ο εισηγητής ανέφερε τον όρο «εποπτεία». Ε, θυμάστε ε, την περίπτωση το Ρουτένιου 106 που ήταν ένα νέφος πάνω από την Ευρώπη και δεν ξέραμε που βρέθηκε αυτό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ε, αυτό το μηχανισμό για να βοηθούμε επιτόπου ε, τους πολίτες και τις ΜΚΟ για να ε, δούμε τι γίνεται στο έδαφος και στο νερό. για τις νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης αλλά δεν θα πρέπει να είναι στα 10 εκατομμύρια, αλλά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, Ρουθένιο 106 ήταν το ραδιενεργό αυτό γνωστοιχείο. Ε, είπατε λοιπόν ότι οι περισσότερες δαπάνες ήταν κάτω των 10 εκατομμύρια ευρώ ε, και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετάει πολύ ε, Μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο ο μηχανισμός για την ασφάλεια, θα πρέπει να επιτακταεί και να καλύπτει ε, όλα τα δεδομένα και όλες τις καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και πρόσβαση στην ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τελίτσκα. On behalf of the ALDE. Από τους φιλελευθέρους. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλό σας απόγευμα. Νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι μολονότι έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολύ μπροστά σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια και τους κανόνες που την διέπουν, καθώς και την τεχνολογία και τις πρακτικές της. Βεβαίως μάθαμε στο παρελθόν ότι κανένα πυρηνικό εργοστάσιο δεν είναι αρκετά μακριά για να μπορεί να μην επηρεάζει μια κοινότητα και την ασφάλειά της. Ε, και αυτός είναι ένας λόγος που θα πρέπει να νοιαστούμε. Από αυτή την άποψη ε, το Άντε συμφωνεί με την πρόταση το σχέδιο της Επιτροπής κατά την άποψή μου είναι ατελές, υπάρχει ανάγκη να συμπληρωθεί τονίζοντας ιδιαίτερα μερικά σημεία. Θα ήθελα να μην επαναλάβω τα ίδια πράγματα, αλλά θα ήθελα να τονίσω μερικά σημεία ακόμα. Καταρχάς, εστιάζεται σωστά η προσοχή, αλλά θα πρέπει να εστιαστεί περαιτέρω το θέμα της μη διάδοσης. Θα πρέπει επίσης να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των διαφόρων χωρών σε ό,τι αφορά τη στάση, την αξιοπιστία των εργαταστάσεων, ε, την, πολιτική, της ε, αξιολογήσεις κινδύνου και περιβάλλοντος που έχουν γίνει. Αλλά σε ό,τι αφορά και ένα πυρηνικό πρόγραμμα Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια πολυσχηδής διαφοροποίηση αυτή που θέλουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε επίσης την προσοχή μας σε θέματα αξιολόγησης, αξιολόγησης κινδύνων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε πρόχειρο ένα σύνολο από μετρήσιμους δείκτες Έχουμε βεβαίως stress test και μία μεθοδολογία, αλλά θα μας απασχολήσουν χώρες που δεν θα έλεγα ότι οι διαδικασίες είναι λιγότερο διαφανείς, αλλά ε, χώρες όπου η αξιολόγηση ε, προσκρούει σε διάφορες δυσκολίες. Θα πρέπει να δούμε τα χρήματα που θα πρέπει να δαπανίσουμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι θα πρέπει να έχουμε μετρήσιμους δείκτες. Σε γενικές γραμμές βρίσκω την πρόταση του εισηγητή, μια πρόταση που θα μπορούσε κατά ένα μεγάλο μέρος να μας βρει σύμφωνους. Θα ήθελα να προσθέσω όμως μερικά σημεία. Δεν νομίζω όμως από ό,τι έχει δείξει η συζήτηση μέχρι τώρα ότι θα υπάρξουν σημαντικές αντιρρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ συνάδελφοι. Ο κύριος Κόλιτσακ από μέρους της ΓΚΟΕ. Κύριε συνάδελφοι, Κύριοι συνάδελφοι, οι συνάδελφοί μου μίλησαν επαρκώς για το θέμα αυτό. Το όλο αυτό θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η συνθήκη της Euratom απαιτεί το κοινό να έχει απόλυτη ενημέρωση σε όλους τους τομείς της διεθνούς συνεργασίας. Τα stress που γίνονται στις διάφορες εγκαταστάσεις θα συμβάλλουν στην ασφάλεια. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ασφάλεια, για προστασία τεχνογνωσίας. Σε ό,τι αφορά τους παρόχους της συγκεκριμένη τεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτευχθεί μια ισορροπία εδώ. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε περιθώρια έμεσου ή άμεσο επηρεασμού των χωρών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν διαφορετική τεχνολογία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις ε, τρίτες χώρες, αλλά πάντοτε με βάση τη συνθήκη της Euratom. Ας αποφύγουμε την εισαγωγή μερικών προκλητικών μέτρων. Η ρήπανση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες. Δεν νομίζω όμως ότι οι χώρες απορρίπτουν την πυρηνική ενέργεια. Δεν νομίζω ότι αυτές που απορρίπτουν χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία ή έχουν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Που θα μπορούσε να προκαλεί ρήπανση ακόμα και σε χώρες που δεν χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια. Τα προγράμματα δράσης είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Παρακαλώ πολύ, ε, ε, όχι πάνω από τέσσερα λεπτά, η κυρία Μέτ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Η κυρία Μέτ. Όχι, εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oh, Well, Α, δεν είναι το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση. Ωραία. Είμαστε απόλυτα ανοιχτοί σε αυτή την αλλαγή. Παρακαλώ. Και πολύ καλές φίλες από το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία. Θα ήθελα. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ σε αυτή τη ε, συζήτηση για το μηχανισμό πυρηνικής ασφάλειας. Διότι συνεργαζόμαστε με αρκετούς ε, συναδέλφους ευρωβουλευτές στενά για το ε, project στο Όστροβιτ, στη Λευκορωσία. Έχουν ήδη γίνει τα stress test εκεί. Και από τη στιγμή που υπάρχουν συστάσεις, νομίζω πως καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Ευρωβουλευτών, που πήγαν στο Μίνσκ και στο Όστροβιτς αυτό ταιριάζει και με όλα αυτά που συζητάμε για τις ε, συνθήκες, ε, δηλαδή για τις προποθέσει αυτού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πυρηνική Ασφάλειας. Η πλευρά της Λευκορωσίας όμως ε, μπλοκάρει οποιαδήποτε συνάντηση και οποιαδήποτε κουβέντα για το Όστροβιτς και το Μίνσκ. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα τη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών που δείχνει πώς πραγματικά κάνουμε τη διαφορά. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την πρωτοβουλία μας, να πάμε στο Μίνσκ για να συζητήσουμε το θέμα του Όστροβιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρμς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκαρίμπα από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. δεν θέλετε να σχολιάσετε. Να με συγχωρείτε, είμαστε από την ε, Γενική Διεύθυνση DevCo. Γι' αυτό και μου έκανε έκπληξη όταν αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ε, ε, λέγεστε Γκαρίμπα. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, μπορείτε λοιπόν να μας συστηθείτε και να τοποθετηθείτε. Ναι, ναι, συγγνώμη για την παρεξήγηση. Λοιπόν, Πασκάλ ονομάζομαι από την ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ, Ανάπτυξη και Διεθνή Συνεργασία, η οποία διαχειρίζεται αυτό το μηχανισμό. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή και το επιτελείο του, διότι είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή πληροφοριών. Η συνεργασία μας ήταν λοιπόν πολύ καλή. Να τοποθετηθώ λοιπόν πάνω σε αυτά που άκουσα. Ως προς το ίδιο το σχέδιο έκθεσης, ένα μόνο σχόλιο έχω για ε, μια τροπολογία στις αιτιολογικές σκέψεις, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη που έχουν προγράμματα πυρηνικής ε, ενέργειας. Ε, έτσι αναφέρει η τροπολογία. Εμείς θεωρούμε πως αυτό δημιουργεί διακρίσεις. γιατί έτσι αποκλείονται κράτη-μέλη τα οποία αυτή τη στιγμή, ε, ενώ είχαν προγράμματα πυρηνικής ενέργειας, προσπαθούν να ε, τα καταργήσουν. Μετά τα stress test. Μην ξεχνάτε πως για την εφαρμογή και την παρακολούθηση ε, υπεύθυνος είναι άλλος οργανισμός, NSREG. Επίσης, ως προς την παρακολούθηση, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα μηχανισμό αποτελεσματικό. Και εάν θέλουμε τρίτες χώρες να υποφεληθούν από τη τεχνογνωσία μας και τον μηχανισμό πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους. Όμως αυτό πρέπει να γίνει δια της διπλωματικής οδού και όχι μέσω ερεσιμότητας όπως αναφέρεται έτσι με πολύ ευθύ τρόπο στο κείμενο. Τέλος, η αιρεσιμότητα που ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι είναι κάτι των ενδιαφέρον, όμως αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο επί τόπου, μόνο κατόπιν των ε, διμερών συζητήσεων με τα κράτη-μέλη που ε, θα ε, θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουρούτσεφ έχει το λόγο, εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις πολύ καλές προτάσεις τους, τα σχόλιά τους πάνω στο σχέδιο έκθεσης. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη μη διάδοση των ε, πυρηνικών όπλων και την ε, πυρηνική ασφάλεια προς τρίτα κράτη είναι πάρα πολύ σημαντική. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Και θα ήθελα να επαναλάβω πως η νομοθεσία αυτή προκύπτει από τη συνθήκη Ευρατόμ. Ας μην συγχαίουμε λοιπόν τις ε, διαδικασίες. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία, διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε δυσάρεστα αποτελέσματα αν ανακατέψουμε την νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. 7 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. 21 Νοεμβρίου θα ε, τις εξετάσουμε. 3 Δεκεμβρίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή και τώρα θα περάσουμε αμέσως στο σημείο 6, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τρία σημεία έχουμε να ψηφίσουμε. Όχι απαραίτητα ηλεκτρονικά, Ξεκινάμε σε τρία λεπτά. It's a great time for me. Yes. Sorry. Good afternoon once again. Καλησπέρα σας λοιπόν ξανά. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Δοκιμαστική ψηφοφορία καταρχάς. Έχετε όλοι τις κάρτες. Υπέροχα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Α, και εγώ πρέπει να ψηφίσω. Λοιπόν, 38. 67 μέλη έχει η Επιτροπή μας. 39. Δεν σας αρέσει η ψηφοφορία της Επιτροπής μας. 40. Τι να κάνουμε, πέρασε. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, λειτουργούν όλα τα συστήματα. Θα περάσουμε στο σχέδιο έκθεσης. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Invest EU. EFCI. Κύριος Σον Κέλλη, ο εισηγητής. Ξεκινάμε. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 170. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε και αυτή ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική τροπολογία α. Πέρας. Εγκρίνεται. 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ταυτόσημη με την 181. Τις ψηφίσαμε και τις δύο. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.15 υπέρ κατά αποχές γκρι... απορρίπτεται. 216 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε τη 216. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε. 260. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 285 και 287 μαζί υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δύο τροπολογίες. 285-287. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτονται. Άλλες δύο, 288-289, υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται και αυτές. Συμβαστική 6, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνατε. Συμβαστική 7, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνατε. 314. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την 314. Πέρας. Εγκρίνεται. 315 και 316. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 317. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. 317. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άλλες 2, 318 και 19. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 350. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 367 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 369 υπέρ κατά Έλεγχο. Την 369 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 370 και 38 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 372 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 374 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 375 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 376 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 377 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 433 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερις τροπολογίες 462, 63, 64, 65 υπέρ κατά. Ας τις ελέγξουμε. Τέσσερις λοιπόν. Ταυτόσιμες. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίνεται, γιατί κανείς δεν λέει το αντίθετο. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 53 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 56 υπέρ κατά απορρίπτεται 57 και 1 μαζί Θέλετε να αλλάξουμε την 56. Πολύ ωραία. Καλή ιδέα. 56 λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα, απορρίπτεται πιο έντονα από ό,τι πίστευα. 57 και 1 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. 57 και 1 μαζί. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85. Υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 85. 85 πέρας ψηφορίας Εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 102. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά έλεγχος 124. Πέρας εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά. Ελέγχουμε την 135. Πέρας. Εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 και 159 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Καλύτερα να είμαστε σίγουροι. Πέρας. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση φυσικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι νομή οδήγηση ευρωπαϊκές μεταφορές. μεταφορέ. εισηγητής είναι ο συναδελφός μας και αντιπρόεδρο επιτροπής μας, κύριος Χένκελ, ο οποίος ζητεί συγγνώμη για την απουσία του και θέλει ε, να σας ευχαριστήσει διαστόματος μου όλους τους γιώδεις και ε, τη γραμματεία. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να φτάσει στις Βρυξέλλες σήμερα εγκαίρος. Γι' αυτό μου έστειλε αυτή την επιστολή να σας τα πω εγώ. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Σχέδιο γνωμοδότησης αυτόνομη οδήγηση ευρωπαϊκές μεταφορές του Hans Olaf Henkel. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 30 το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ φωνές από κάτω. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συγγνώμη, εγκρίθηκε. Ζητώ συγγνώμη. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ. Κατά αποχές, και ε, αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές. Ας την ελέγξουμε για καλοκιά κακό, είναι 53 πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν σηκώνεται χέρια. Ας την ελέγξουμε και πάλι λοιπόν. Πέρας. Απερίφθη. Κάτι είχα υποπτευτεί. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 69 ψηφίζουμε. παρακαλώ. Εγκρίθηκε. Η συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 71, το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71, το δεύτερο τμήμα του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 72. Η Γκου έχει ζητήσει εδώ ονομαστική κλίση. Και στην Επιτροπή μας θα πρέπει τουλάχιστον 14 μέλη να δεχτούν μια τέτοια πρόταση για να τέθει σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση η τροπολογία. Σας ερωτώ λοιπόν, θέλετε να ψηφίσουμε την τροπολογία 72 με ονομαστική κλίση υπέρ παρακαλώ μια τέτοια πρόταση. Μάλιστα, ωραία. Είναι πάνω από 14. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση λοιπόν την τροπολογία 72. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 76 υπέρ κατά έλεγχος. Παρακαλώ να τσεκάρουμε την 76. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται συμβαστική δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, την τέσσερα η τέσσερα ήτανε ψηφίσαμε την τέσσερα προηγουμένως η τροπολογία 4 η επόμενη θα είναι η 5 Ξανά. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε. Τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ορίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 14. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα και τελειώνει εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον απόντα εισηγητή μας. Προχωρούμε λοιπόν στο σχέδιο έκθεσης για τη τεχνολογία blockchain, μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική. Εισηγητής είναι ο κύριος Μπουσόη. κύριε Μπουσόη, ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου. Και ψηφίζουμε ευθύ αμέσω. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά έλεγχος. Παρακαλώ να παληθεύσουμε την 23 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτή τη φορά. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά ας το επαληθεύσουμε αυτό παρακαλώ 48 πέρας απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές και αυτό θέλει επαλήθευση μάλλον το 49 ψηφίζουμε την τροπολογία 49 πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα, η τελική παρακαλώ, αρχίζει τώρα. And I close. Και τελειώνει ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη υποστήριξη. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά για την έκθεσή σας. Σχέδιο γνωμοδότηση ήταν, για την γνωμοδότησή σας. Well, leaving, incredible. let us start then. Let us start. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε αγαπητοί φίλοι. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Mrs. Toy is coming in a second. The rapporteur. Ah, okay. Good. The most important lady is coming. That's important. Great. Okay. Uh, point number Λοιπόν, στο σημείο 9 είμαστε θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Γνωμοδότηση είναι η δική μας και είμαστε ε, αρμόδιοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα. Και ξέρουμε ότι έχουν κατατεθεί 188 τροπολογίες σε αυτή τη νομοθετική γνωμοδότηση. Κοιτάξτε, διαδικαστικά θέλω να πω το εξής. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα, με πέντε συναρμόδιες επιτροπές που έχουν κάθε μία αποκλειστικές αρμοδιότητες και οι τροπολογίες για τα άρθρα, τα παραρτήματα, τις αιτιολογικές σκέψεις που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων επιτροπών πλην της Ήτρες, στο μέλλον δεν θα ψηφίζονται. Γιατί αποκλειστικότητα σημαίνει αποκλειστικότητα. Άρα, για μας αυτό τι σημαίνει. Πάρα πολύ καλά νέα. Διότι αποτελεί εγγύηση ε, ότι η δική μας επιτροπή θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για το σκέλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κανείς δεν θα μπορέσει να ψηφίσει σε άλλη επιτροπή τροπολογίες, μόνο εμείς. Πολύ καλά νέα. Η κυρία Πατρίτσια Τόια, συνάδελφος, αντιπρόεδρος, είναι αρμόδια για το θέμα αυτό και της δίνω μέσω στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε σήμερα να ξεκινήσουμε μία συζήτηση που θα μας προχωρήσει λίγο στην εξέταση αυτού του θέματος που όπως είπες και εσύ παρουσιάζει ορισμένες πολυπλοκότητες γιατί παρεμβαίνουν διάφορες επιτροπές. Το πρόγραμμα αυτό το συλλάβαμε έτσι γιατί δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να τα βάλουμε όλα μαζί. Υπάρχει ο κίνδυνος, το δικό μας κομμάτι, να είναι όχι περιθωριακό αλλά λιγότερο σημαντικό. Είναι καλή η ιδέα που παρέθεσες κανένας ε, δεν θα μπορέσει να ασχοληθεί με τις ε, ΜΜΕ, αλλά το αντίθετο του ε, νομίσματος είναι ότι εμείς θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό το πεδίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους για τη συμβολή τους, όχι μόνο σε επίπεδο τροπολογιών, αλλά και με τις συζητήσεις που είχαν οι συνεργάτες μας σε δύο τεχνικές συζητήσεις που θα μας βοηθήσουν αύριο στις συναντήσεις με τους συζητητές και τους χειώδεις ηγητές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για τη δουλειά που έκαναν δουλειά που αφορούσε και τι τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα να δεκτώ όσο γίνεται περισσότερες τροπολογίες, γιατί όπως κάναμε στην πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή υπάρχει μεγάλη σύγκριση, σύγκληση σε ό,τι αφορά το στόχο των ΜΜΕ και πιστεύω ότι η συμβολή όλων μας θα εμπλουτίσει το κείμενο. Το κείμενο. Θα ήθελα καταρχά να υπογραμμίσω ένα πρώτο σημείο που αφορά και τις τροπολογίες αλλά και την διατύπωση. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλες οι ομάδες απέδωσαν σημασία στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλοι επιθυμούμε μία ανάπτυξη, δεν θέλουμε να διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει. Θα γίνουν λοιπόν δεκτές όλες τις τροπολογίες που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το θέμα της βιωσιμότητας, ορισμένες ομάδες επιμένουν περισσότερο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, άλλες ομάδες πιστεύουν ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτός ο όρος, κατά την άποψή μου, η ε, βιωσιμότητα είναι ένας πυλώνα και αυτό μας το δείχνουν τα γεγονότα. Και υπάρχει και το θέμα της ε, διαχείρισης. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχει στόχο την τον τον εσοδεύσει της ε, ΜΜΕ στην ψηφιακή μετάβαση η οποία έχει βεβαίως και μερικά θετικά σημεία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Βεβαίως υπάρχει και ένας άλλος στόχος που αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Θέλουμε να υπάρξει ένα ανταγωνιστικό και δυναμικό σύστημα προκειμένου να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Σε ό,τι αφορά το θέμα ε, οργάνωσης θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό και ένα άλλο κριτήριο που θα απασχολήσει τους ε, συναδέλφους την υποστήριξη των ΜΜΕ σε ό,τι αφορά την ε, προετοιμασία των κατάλληλων μάνατζερ. Πολλές φορές το προϊόν που έχουν είναι καλό, αλλά λείπει μια καλή διαχείριση. Κάτι άλλο επί του οποίου συμφώνησαν οι ε, ομάδες είναι ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί το πρόγραμμα COSME. Το ένα είναι European Enterprises ε, ε, Network και το άλλο αφορά την αξιοποίηση του προγράμματος Εράσμους που θα πρέπει να επανέλθει στον αρχικό του, στο αρχικό του επίπεδο και εδώ θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη αν θα ε, αφορά τους νέους επιχειρηματίες ή ε, ε, θα πρέπει, θα πρέπει να αφορά γενικά τους επιχειρηματίες νέους ή λιγότερο νέους. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στο ακαθόδε θέμα των δικτών για την ετήσια έκθεση. Η Επιτροπή παρουσίασε μερικούς δείκτες Μερικοί από εμά μέλη του Κοινοβουλίου, εμπλούτησαν τους δύο δείκτες της Επιτροπής. Εδώ θα πρέπει, πιστεύω, να κάνουμε μία επιλογή, να διασώσουμε μερικά βασικά σημεία που προτείνεται, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και κάπως να περιοριστούμε εμείς. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω αφορούν δύο σημεία που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, αλλά μερικοί είπαν ότι είναι υπέρ. Θα πρέπει μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων να λάβουμε υπόψη μας και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν στόχο να, την κερδοφορία, αλλά την δημιουργία θέσεων εργασίας. Ή αυτές είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Έχουν δηλαδή μια διαφορετική, ε, βλέπουν το θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Οι κοινωνικές λοιπόν επιχειρήσεις δεν αποσκοπούν στην κερδοφορία αλλά στη δημιουργία θέσεων εργασία και έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρο σε αυτό το πρόγραμμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ένα τελευταίο σημείο, αύριο θα πρέπει να ε, διευκρινίσουμε το θέμα των δικτύων επιχειρήσεων, το Enterprises Network. Θα πρέπει να γίνουμε περισσότερο ε, ακριβείς. Δεν είναι ένα απλό κλάστερ, είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων επιχειρήσεων ε, που παρέχουν υπηρεσίες ή που εργάζονται στον ε, τομέα μεταποίησης. Είναι ένα είδος κονσόρτσιουμ ε, ε, κοινοπραξίας επιχειρήσεων αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι μάλλον μια ε, καινοτομία, η δημιουργία δηλαδή ε, αυτών των ε, σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας αλυσίδας αξίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και λυπάμαι που ξεπεράσα το χρόνο που μου είχατε δώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ο κύριος Ρούμπικ ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρου ε, του ΕΛΚ θα μυρίσει αργότερα. Ο κύριος Τελίσκα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. Ε, νομίζω πως είχαμε μια καλή συνεργασία. Οι τροπολογίες μου και της ομάδας μου ε, έγιναν αποδεκτές, συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο γνωμοδότησης. Τώρα αυτό που απομένει είναι ορισμένες ε, λεπτομέρειες, διευκρινήσεις ε, λεπτομέρειες, τα παραρτήματα για παράδειγμα βρίσκω κάποια περιτά σημεία Από την άλλη δεν βλέπω να αναφέρεται η στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτά είναι μικροπράγματα που πιστεύω πως θα λύσουμε ε, στην πορεία. Αύριο είναι η πρώτη συνάντηση, γι' αυτό λοιπόν ε, θα απαντήσω έτσι στην έμεση ερώτηση της κυρία Τόγια που έκανε στο τέλος για τα σημαντικά θέματα, καταρχάς ε, για το Εράσμους. Να πω πως έχει απόλυτο δίκιο τώρα για το πόσο, για θεωρείται κάποιος νέος και ποιες είναι αυτές οι ηλικίε, αυτό είναι κάτι άλλο. Είχα κάποιες αμφιβολίες για την ε, χρήση του ίδιου του Εράσμους. Όταν είμαι επιχειρηματίας δεν μπορώ να λείψω για πάρα πολύ καιρό από την επιχείρησή μου, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως μία βραχία περίοδος θα ήταν πιο λογική. Μπορώ να συμφωνήσω ε, επί της ουσίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, είναι μία καλή ιδέα θα έλεγα. Ε, για τα δίκτυα, τα επιχειρηματικά δίκτυα. Νομίζω πως ο δικός μας ρόλος έχει να κάνει με τη στήριξη της δημιουργίας και της διαχείρισης αυτών των δικτύων. Όμως, εδώ πρέπει να διευκρινιστούν κάποιες λεπτομέρειες, σε μικρά πράγματα. Είμαι σίγουρος πως στο τέλος θα, θα καταφέρουμε πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε ένα καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Και εδώ να πω πως εκτιμώ τις προσπάθειες της εισηγήτριας να συμπεριλάβει τις τροπολογίες μας στο σχέδιο γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μέτς έχει το λόγο εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Δεν θα πω πολλά σήμερα. Καλά πάει η δουλειά, έχουμε καταθέσει τροπολογίες για τη βιωσιμότητα, την ε, ε, αποδοτικότητα των πόρων. Πιστεύουμε πως αυτά πάνε χέρι με χέρι με την ανταγωνιστικότητα. Επίσης παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι κάπως ασαφής η διατύπωση, ιδιαίτερα σε σχέση με τα διάφορα προγράμματα και σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να σας πω ότι στην COSME Αναφέρθηκαν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, ε, κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες ε, κατάρτιση σεμιναρίων για την επιχειρηματικότητα και άλλα ε, στοιχεία που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν, δηλαδή πώς μπορούν να μειώσουν το διοικητικό φόρτο κτλ. Εκτιμούμε πολύ την αναφορά στον συμβουλευτικό κόμπο, αυτό το Advisory Hub, στο πλαίσιο του InvestEU. Επίσης, νομίζω πως η μοναπευθυντική θηρίδα θα ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που ε, συμπεριέλαβε τις ε, τροπολογίες μας και ε, τις εξέτασε. Σας ευχαριστώ πολύ. εκ μέρους της ΓΚΟΥ, η κυρία Λόπες Περμέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της. Νομίζω ότι οι συμβαστικές της προτάσεις ε, μπορούν ε, να μας βρουν ε, σύμφωνους ευρεία συνέρευση σε αυτό το θέμα που δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι δικές μας τροπολογίες θέλησαν να διορθώσουν λίγο τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η εσωτερική ενιαία αγορά στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Μπαίνω στην ουσία του θέματος από τη μια συμφωνούμε με τη συμμετοχή πολιτών και καταναλωτών στη διαδικασία ε, ενημέρωσης και λήψης απόφασης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως προϋπόθεση ε, για να έχει κανείς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα COSME ε, πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση αυτή η προοπτική, αλλά δεν θα πρέπει να μείνει μόνο στο διακηρυκτικό ε, στάδιο και στις προθέσεις. Θέλουμε να είναι πραγματικά λειτουργική και να εφαρμοστεί και να χωρούν και νέες μορφές ε, επιχειρήσεων. Ανέφερε η συγγήτρια τι γίνεται με τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα πρέπει να εθαρρυθεί η συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, και με τα ιδρύματα που παράγουν γνώση όπως είναι τα επιστημονικά, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κτλ. Χρειάζεται ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον δυναμικό, κοινωνικά υπεύθυνο. Όλα αυτά ε, δεν γίνονται με αυτοσχεδιασμούς και ούτε μπορούν φυσικά να αφαιθούν στις δυνάμεις της αγοράς, γιατί οι δυνάμεις αγοράς πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση λειτουργούν. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε χώρο σε αυτές τις κοινωνικές εταιρείες, να ε, τις προβάλλουμε, να γίνουν γνωστές και να προωθήσουμε την ε, ανάπτυξή τους και την μεγέθησή τους. Έχει έρθει ε, η ώρα για την κοινωνική ε, Ευρώπη και ε, για τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη λήψη αποφάσεων στις εταιρείε και στην ενημέρωση, τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή κτλ. Όλα αυτά τα θέματα είναι μεγάλου βεληνικούς. Ελπίζουμε να καταλήξουμε και εμείς σε μια ευρύτατη συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο ε, κύριος Κόχλιτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Τρία πράγματα έχω να πω μόνο για το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τους συνεταιρισμούς, έτσι, που θα χρειαστούν και αυτή τη στήριξή μας οπωσδήποτε. Δεύτερον, οι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, χρειάζονται υποστήριξη και να αναφέρονται ρητά. Και τρίτον, τα λεγόμενα ε, εκολαπτήρια, incubators ε, των μικρών πολυ... και νεοφυών επιχειρήσεων ε, και να γίνει και μια αναφορά στο πρόγραμμα Έρασμος, γιατί ο Έρασμος θα πρέπει να ε, ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των νέων. Ευχαριστώ. Από την DG Grow, ο κύριος Γκέτ Σμίτς, έχετε το λόγο. Um, thank you everybody. Uh, the Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της ενίας αγοράς, αλλά και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη θετική σας στάση στο πρόγραμμα αυτό και την πρόοδο που έχει σημειωθεί καθώς και την επιθυμία σας για ε, ταχεία ολοκλήρωση του φακέλου. Ε, ένα σχολείο για το Εράσμους και για τους ε, νέους. Ε, αναφέρεται η πρόταση στην ηλικία της επιχείρησης και όχι του επιχειρηματία. Είναι δηλαδή για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο πίσω στην εισηγήτρια, κυρία Τόγια, για τα καταληκτικά σχόλια. Βεβαίως με το Ρούμπικα θα έχουμε μία διμερή ανταλλαγή απόψεων. Σε κάθε περίπτωση είχαμε την ευκαιρία ήδη να το συζητήσουμε το θέμα. Θα είναι επικοδομητική αυτή η συζήτηση, όπως επικοδομητικές υπήρξαν όλες οι παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλες οι υποθέσεις για να γίνει μία σωστή δουλειά αύριο θα συναντηθούμε, δεν υπάρχουν πάρα πολλές ε, αντιθέσεις, απλά και μόνο θα πρέπει να συμφωνήσουμε περιορισμένο σημείων. Ε, νομίζω ότι όλες οι ιδέες είναι χρήσιμες για αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει να το διευρύνουμε, θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Ε, θα γίνουν δεκτά ε, όλα όσα χρησιμεύουν στο να βελτιώσουν αυτό το πρόγραμμα. Συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και πράγματα που δεν είναι ε, σημαντικά σήμερα, αλλά θα γίνουν σημαντικά αύριο. Θα βρούμε κάποιο τρόπο να τα εντάξουμε και ε, να το ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Uh, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία στο ΙΤΕ 3 Δεκεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου και ψηφοφορία στην ΕΜΚΟ 22 Ιανουαρίου του 2019. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Δημιουργία ενό ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Ο στόχος της πρότασης είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που προσπαθούν να κλείσουν τις πυρηνικές ε, εγκαταστάσεις. Αυτή η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 203 της συνθήκης Euratom. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο θα υιοθετήσει αυτόν τον κανονισμό αφού ζητεί την άποψη του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς βεβαίως να έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει την γνωμοδότησή του. Ο ο εισηγητής είναι ο Πίτερ Κορουμπάσεβ. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τις βασικές ιδέες που υπέβαλαν οι πολιτικές ομάδες. Με βάση τις τροπολογίες τους θα έλεγα ότι η ομάδα των Πρασίνων και η ομάδα της Γκουε είναι υπέρ μιας πιο ενεργής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προγράμματα παρεπουλισμού. Από το 50 θέλουν να περάσουμε στο 60%. Οι βασικές διαχωριστικές γραμμές σε αυτή την ε, έκθεση έχουν να κάνουν με την πρόταση της ε, ΓΚΟΕ ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα ποσοστά χρηματοδότησης. Η Επιτροπή επίσης προτείνει να μειωθούν οι δεσμεύσεις της ή ένα μέρος αυτών. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 60% ε, στο είναι 63%. Η Επιτροπή προτείνει οι δεσμεύσεις να μειωθούν στο 50%. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σχετικό. Ο κύριος Λάγκεν ανέφερε ότι ότι όταν μια χώρα παίρνει την απόφαση να παροπλήσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο θα πρέπει να έχει και τους απαιτούμενους πόρους για τέτοιο πρόγραμμα. Ούτε η Βουλγαρία, ούτε η Σλοβακία, ούτε η Λιθουανία δεν πήραν την απόφαση να παροπλήσουν τα πυρηνικά εργοστάσια τους. Η απόφαση αυτή υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προϋπόθεση για αυτές τις χώρες ήταν να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι συνάδελφοι προβληματίζονται γιατί πιστεύουν ότι η οικονομική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο στο μέλλον. Δεν νομίζω όμως ότι είναι βάσιμες οι ανησυχίες τους ε, γιατί η ο παραπλισμός στην Πόχουνίτσα και στο Κοσλοντούι ήταν απαραίτητη προϋπόθεση ένταξη των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα συνάδελφο από την ομάδα ECR έθεσε το θέμα των τρίτων χωρών παραπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες. Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί μία ομάδα στο κοινό ερευνητικό κέντρο ένα κέντρο το οποίο θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που έχουμε από τα προγράμματα παροπλισμού. Τα προγράμματα αυτά θα είναι χρήσιμα όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για όλο τον κόσμο. Τα προγράμματα παροπλισμού δεν θα πρέπει να είναι όμοιροι της πολιτικής ε, ε, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος έχει εμπειρία παροπλισμού θα πρέπει να τη μοιραστεί και με άλλες χώρες για λόγους ασφαλείας που αφορούν και τη χώρα αυτή και όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα ανώτατο κατόφλι για τη συμμετοχή της Επιτροπής. Αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι 50%. Εγώ θα πρότεινα ένα ελάχιστο εδώ, ένα ελάχιστο κατόφλι για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια σαφή δέσμευση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα προεπαιτούμενα τα έχουν αναφερθεί από τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά τους πράσινους και την ομάδα Γκουε. Υπάρχουν μερικές διαφορές ε, με το Ελκ και κυρίω με τον κύριο Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάντ, έχετε το λόγο. Σε γενικές γραμμές ε, θα μπορούσα να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση των συναδέλφων ε, για τις τροπολογίες. Ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες που αφορούν την έκτακτη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα παροπλισμού. Μιλάμε για το Κοσλοντούι, την Μποχονίτσα και μετά για την Ιγναλίνα. Μιλάμε για κατεξαίρεση περιπτώσεις, δεν μιλάμε για τον κανόνα. Ο κανόνας ε, στην ομάδα μου αλλά και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι χώρες, μέλη και η πυρηνική βιομηχανία είναι υπεύθυνοι για τον παροπλισμό, για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Μπορώ να καταλάβω όμως ότι οι συνάδελφοι θέλουν να υπογραμμιστεί περαιτέρω αυτό. Σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση, συμφωνώ με τον κύριο Κομπάτσεφ, οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει ως προς το σημείο αυτό για την Ποχονίτσα και τον Κοσλοντούι αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή το, το, το κατόφλι συγχρηματοδότηση της ε, Ένωσης θα πρέπει να συμφωνήσει με την πρακτική του προγράμματος του προκατόχου. Δηλαδή θα, οι χώρες μέλη θα, ε, θα, πρέπει ε, ε, να μπορούμε να βασιστούμε όταν μιλάμε για το θέμα ε, της συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Γουπάτσεφ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Κύριος Λάγκεν από την ομάδα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί ψήφισα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, γι' αυτό λοιπόν καθυστέρησα να έρθω. Ο συνάδελφος Κουρουμπάτσεφ έχει διατυπώσει μία πρόταση η οποία σε πολλά σημεία μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμάς, αλλά Υπάρχουν κάποιοι κανόνες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση, στους οποίους θα θέλαμε να κάνουμε κάποια σχόλια. Προτείνει λοιπόν ο εισηγητή αντί για ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν ελάχιστο, ένα ελάχιστο ποσοστό 60%. Αυτό ε, είναι αντίθετο σε όλα τα άλλα προγράμματα ε, συγχρηματοδότησης, τα οποία έχουν ανώτατο ε, συντελεστή. Αυτό, ε, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι με μικροποσά, είναι τεράστια ποσά και πρέπει να τηρήσουμε τους ε, κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να πάρουμε την πρόταση αυτή του εισηγητή στα σοβαρά. Μπορούμε απλά να εκφέρουμε λοιπόν αυτή την άποψη. Μετά, ε, οι τροπολογίες 5 και 6, όπου ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιάμεση αξιολόγηση, προτείνουμε να διαγραφούν για να εξετάσουμε εάν μπορούν οι πόροι να διατεθούν ε, με διαφορετικό τρόπο. Η πρόταση της Επιτροπής ε, μου φαίνεται αρκετά πιστική. Ο παροπλισμός των εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία έχει προχωρήσει αρκετά. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω πως είναι δυνατόν στην ενδιάμεση εξελόγηση του που, που να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την εξελόγηση και να διατεθούν αλλού οι πόροι, να αλλάξουν τα ποσοστά χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πως είναι προς το συμφέρον όλων ε, και από όλε τις ε, πλευρέ να γίνει γρήγορα παροπλισμό των ε, εργοστασίων αυτών. Και για περιβαλλοντικού λόγους και για ερευνητικού λόγους. Ο κύριος Κουρμπάτσεφ λοιπόν έχει υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Η ομάδα μου έχει υποβάλει μία τροπολογία, 21, τροπολογία 21 για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, της κυρίας Γκροστέ, την οποία και φυσικά θα ε, υπερψηφίσω. Οι άλλες μας φαίνονται εντάξει, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, παροπλισμός, ε, εδώ θα είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για τον παροπλισμό. υπάρχουν κάποιες τροπολογίες από την ομάδα ECR με τις οποίες επίσης δεν έχουμε κάποιο θέμα και οι τροπολογίες της κυρίας Χάρμς και Σιλουάγκαμ από την ε, Γκουε Θέλουν επίσης ε, ποσοστό 60% συγχρηματοδότησης. Υπάρχουν εδώ διαφορές, ε, αλλά νομίζω πως ε, δεν χρειάζεται να γίνουν συναντήσεις και οδόν. Μπορούμε απλά να καταρτήσουμε έναν κατάλογο ψηφοφορίας και να τον ψηφίσουμε, διότι δεν μπορούμε να βρούμε κάποια αποδεκτή συμβαστική λύση όταν υπάρχουν τόσο διαφορετικές αποκλήσεις απόψεων από τις διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμβιβαστούμε. Όλοι έχουμε τις γραμμές μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας παρακαλώ να ψηφίσουμε στο τέλος ε, του Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Ο κύριος Κόχλιτσακ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι ο κύριος Λάγκεν, όπως πάντα, είναι συνεπής στα λόγια του. Συμφωνώ μαζί του σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ή τη διατύπωση μάλλον, ε, δηλαδή για τα μέγιστα ή τα ελάχιστα ποσοστά της ε, συγχρηματοδότησης, γιατί όχι ας τα ψηφίσουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα ελάχιστο ποσοστό και σε ένα μέγιστο ποσοστό, αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβασμό. Σίγουρα το 50 δεν ισούται με το 60, ο κύριος Λάγκεν το κατέστησε σαφές. Κύριε Κορουμπάτσεφ, συμφωνώ μαζί σας με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν ε, θέλουμε να κάνουμε λόγο για προηγούμενο, για δημιουργία προηγούμενου που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν και οι συνθήκες προσχώρησης και πρέπει να εξετάσουμε το αν ισχύουν ακόμα οι διατάξεις των συνθήκων αυτών ή όχι. Πιστεύω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε γι' αυτό, αν θα αποτελέσει δηλαδή προηγούμενο για το μέλλον, για την περίπτωση προσχώρησης ε, χωρών που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε αν είναι ε, δεσμευτικές ή όχι συνθήκες. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, 50%, 60% το 55% είναι συμβιβασμός. Το ξέρω, το ξέρω και αστείευομαι. Εννοείται. Φυσικά και έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, τον κύριο Μάσιμο Γκαρίμπα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση. Και επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι η πυρηνική ασφάλεια είναι από τις κυριότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ πρέπει να δούμε ότι ο παροπλισμός των εγκαταστάσεων αυτών είναι και μία ένδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες αυτές και μάλιστα είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις στον παροπλισμό τους. Η όλη συζήτηση για τα ανώτατα όρια, για τα κατόφλια για το ποια θα πρέπει να είναι δηλαδή τα όρια, ποιο θα πρέπει να είναι το επίπεδο της αλληλεγγύης. Γι' αυτά έχω να πω τα εξή. Τα επίπεδα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν με τις οικονομικές ανάγκες ε, του παροπλισμού των ε, εργοστασίων αυτών. Να σας υπενθυμίσω ότι οι εγκαταστάσεις των Μποχούνιτσε θα παροπλιστούν πλήρως μέχρι το 2025 και οι εγκαταστάσεις στο Κοσλοντούι μέχρι το 2030. Η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης ήταν κάτι που πάντα υπήρχε στα προγράμματα αυτά. Αυτό δείχνει την ε, δέσμευση των κρατών μελών ως προς τον παροπλισμό. Τώρα, οι ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι συνάδελφοι είναι φυσικά σωστές και εδώ έχω να πω ότι η γνώση που έχουμε αποκτήσει θα βοηθήσει έτσι ώστε τα χρήματα των φορολογούμενων που θα διατεθούν για τον παραπλησμό να διατεθούν σωστά. Σίγουρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας με τους ε, υπόλοιπους ε, αρμόδιους φορείς θα φροντίσουν για την διάδοση των πληροφοριών αυτών και τη διάδοση της γνώσης. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα δώσω τώρα τον λόγο πίσω στον εισηγητή κύριο Κουρουμπάτσεφ. Έτσι ώστε να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να τονίσω ότι στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Σλοβακίας οι δύο αυτές χώρες είναι ένα υπόδειγμα σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό παροπλισμό. Στη Σλοβακία θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το 2025 και στην Βουλγαρία προβλέπεται και το 2030. Τώρα ως προς τα ποσά δεν είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Για τα επόμενα 7 χρόνια προβλέπεται ένα κόστος 27 εκατομμυρίων ευρώ, 9 δηλαδή εκατομμύρια το χρόνο. Για την ε, Σλοβακία 8 εκατομμύρια το χρόνο. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε προβάλει εξευτελιστικές απαιτήσει κατά τη διάρκεια των συνομιλίων ε, προσχώρησης, ο παροπλισμός αυτών των πυρηνικών εργοστασιών θα είχε καθυστερήσει και θα δημιουργούσε έσοδα 400 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Αυτά δεν συγκρίνονται καν με το ποσό που εισπράττουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 9 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και μάλιστα τώρα συζητάμε αναρωτιέται το ενδεχόμενο να μειωθεί αυτό το ποσό στα 8 ή ακόμα και στα 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είμαι υπέρ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών, την πρόταση δηλαδή των συναδέλφων του ΕΛΚ και των ε, φιλελευθέρων. Ο παροπλισμός, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σε επίπεδο κοινών ομάδων εργασίας ή του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Έτσι ώστε η εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά τον παροπλισμό να συγκεντρωθεί και να χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Θα είναι πολύ σημαντικό μια που ο παροπλισμός θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα της Ένωσης στο μέλλον. Και θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό για τα ανώτατα ή τα ελάχιστα όρια. Αυτό νομίζω θα, θα φανεί και από τη συνάντηση των σκιωδών και μετά θα δούμε πώς θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο κύριο Λάγκεν ζητεί το λόγο για κάποιο σχόλιο συμπραγματικό. Παρακαλώ. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν εναλλακτική λύση θα ήταν η συνέχιση ε, της λειτουργίας. Αυτό το συζητάω, αλλά δεν το προβλέπουν αυτό οι συνθήκες προσχώρησης. Ε, γεγονός είναι ότι ε, απέτησαν τον παροπλισμό με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομική. Ε, δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει ε, τα ενδεχόμενα έσοδα ε, και να τα συμψηφίζει με τα εξοδα παροπλισμου παραπλισμού από ένα κλειστό εργοστάσιο. Είναι πάνω από ένα-δύο δισεκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που έχουν εκταμιευθεί για να κλείσει το εργοστάσιο αυτό. Δηλαδή μην μας λέτε κιόλας ότι ε, είναι διακριτική μεταχείριση εις βάρος της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας που συμφώνησαν ε, στην ε, προσχώρηση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περηφανεύεται κατά τα άλλα ότι είναι υπέρ της μεγάλης ασφάλειας το κάνετε αυτό παντού, το επιβάλλετε και στη Γαλλία, αν σκεφτώ το εργοστάσιο του Φέσενχάιμ. Είναι πάρα πολύ χολή αυτή η επιχειρηματολογία. Να το σκεφτούμε όσο θέλετε, αλλά συμβασμό δεν πρόκειται να βρούμε. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει συνεδρίαση των σκιωδών. Δεν ε, χρειάζεται. Για 21 τροπολογίε τι να την κάνουμε, να συμβαστούμε δεν πρόκειται. Ευχαριστώ. Η απόφαση θα ληφθεί από τον εισηγητή φυσικά τον ίδιο. Κύριε Κόχλητσακ, τι έχετε σχόλιο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε το λόγο τώρα. Ο εισηγητής, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κατά τη δική μου άποψη, είναι απαραίτητη η συνεδρίαση των σχεδόν. Τουλάχιστον μία συνεδρίαση σχεδόν εισηγητών χρειάζεται, πιστεύω. Ακόμα και αν στο τέλος ε, θα καταλήξουμε σε μια απόφαση που λέει ότι δεν χωράει συμβιβασμό. Υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες, λίγες, ε, που με υποστηρίζουν. Μπορεί να υπάρχουν άλλες πολιτικές ομάδες που να υποστηρίζουν την ε, επιχειρηματολογία και το σκεπτικό του κυρίου Λάγκεν. Κατά την προενταξιακή διαδικασία, μας έστειλε τελεσίγραφο σε ορισμένες χώρες για το παροπλισμό των πυρηνικών εργοστασίων. Και η πλευρά που έθεσε αυτό το τελεσίγραφο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει και τη διαδικασία παροπλισμού. Εάν έρχεται μια χώρα και παίρνει την απόφαση να παροπλήσει τα πυρηνικά της εργοστάσια για τον, δια... λόγο, θα πρέπει να αφιερώσει και απαραίτητα χρήματα. Εάν όμως μια χώρα υποχρεώνεται να πάρει αυτή την ε, απόφαση κατά τη διαδικασία των προενταξιακών διαπραγματεύσεων, τότε θα πρέπει εκείνο που επιβάλλει την απόφαση αυτή να αναλάβει ε, το σύνολο της χρηματοδότησης. Τώρα συζητούμε για 9 εκατομμύρια ετησίως για την ε, Βουλγαρία και 8 για τη Σλοβακία. Και σας ανέφερα και την ενέργεια που παράγεται τώρα και θα παραγόταν μάλλον από τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία αν ήταν ε, σε λειτουργία τώρα τα εργοστάσια μας. Και ε, θα ήταν πολύ περισσότεροι ε, τα έσοδα που θα είχαμε από τη δαπάνη. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κ. Σκόχλητσα, στα γερμανικά. Κύριε Λάγκεν, ζητώ συγγνώμη. Όταν υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εδώ, ε, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και σε όλα τα Βαλκάνια δεν βοήθησε καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό είναι πολύ λογική η απέτηση αυτή ή το αίτημα να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λογικό αυτό και εσείς λογικά σκεπτόμενος ε, είστε και πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε. Δέχεστε αυτό το λογικό επιχείρημα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Αν προσπαθήσω τώρα εγώ, Ρομίρ να σκεφτώ και εγώ λογικά, θα έλεγα το εξής. Είναι απαραίτητη η συνεδρίαση των σκιωδών, γιατί δεν μπορεί εδώ να τελειώσει η συζήτηση αυτή. Αν δεν συνεδριάζουν οι σκιώδεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε καθόλου διότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λέει ο κύριος Λάγκεν είναι 21 τροπολογίες. Τι θέλουμε ολόκληρη συνεδρίαση. Ε, ε, ε, Τίστε και κανένα κουμπάκι γιατί μιλάτε εκτός μικροφώνου. Μα δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε συνεδρίαση σκιωδών. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε τις 21 τροπολογίες, 21. Στην κανονική συνεδρίαση. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Okay, okay. Our, our meeting is absolutely official. Βεβαίω είναι επίσημη η συνεδρίασή μας πάντα, αλλά και σκιώδει ε, εισηγητέ συνεδριάζουν. Αυτό εξαρτάται από τον εισηγητή. Ω συνήθως στην Επιτροπή μας αυτό γίνεται, δεν έχουμε άλλους κανόνες. Καταλαβαίνω ότι και εσεί λέτε ότι δεν χρειάζεται συνεδρίαση των σκιωδών για 21 τροπολογίε, αλλά οι απόψει διήστανται. Το χέρι σα είναι. Λοιπόν, εντάξει όλα είναι στο χέρι σας. Λοιπόν, πάμε. Προχωρούμε. Ο κύριος Κορουμπάσεφ. Θα ήθελα παρακαλώ να πω το εξής. Ε, καλό καλώ όλους τους συναδέλφους σκιώδης στη συνεδρίαση των σκιωδών την άλλη εβδομάδα. Και όποιος θέλει, καλώς να ορίσει. Όποιος δεν θέλει ή δεν το θεωρεί σκόπιμο ή δεν ε, θέλει, ε, είναι επίση ελεύθερος να μην έρθει. Θα προγραμματίσω στο Στρασβούργο συνεδρίαση των σκιωδών και πάρτε τις αποφάσεις σας παρακαλώ. Αν θέλετε να έρθετε και όποιο δεν θέλει, καλώ και αυτό. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ε, στις 3 ε, Δεκεμβρίου ε, στην Επιτροπή μας, λέει ο Πρόεδρος. Και προχωρούμε στο σημείο 11. Αντίστοιχο σημείο. Πρώτα κανονισμό του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού Ιγναλίνα στη Λιθουανία. Όπως γνωρίζετε, νομική βάση για αυτό το θέμα δεν προβλέπει, δεν απαιτεί μάλλον διαβούλευση του Κοινοβουλίου, αλλά το Συμβούλιο αποφάσισε να μας ζητήσει τη γνώμη μας. Ε, όπως στην περίπτωση της Σλοβακίας και της ε, Ρουμανίας και Βουλγαρίας προηγουμένως, συγγνώμη. και προτείνει τώρα για το πυρηνικό σταθμό Ιγναλίνα ε, στη Λιθουανία το πρόγραμμα παροπλισμού και προϋπολογισμό φυσικά για την περίοδο 2021-2027. Η συγκήτρια είναι η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς, η οποία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να κάνω μια εισαγωγική παρατήρηση ε, που συνδέεται με την προηγούμενη συζήτηση Κουρουμπάσεφ Κόχλιτσεκ και Λάγκεν. Ε, είναι τρία τα πυρηνικά εργοστάσια που συζητούμε σε δύο εκθέσεις, Ιγναλίνα, Μποχουνίτσα και Κόσλοντουή. Και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των προενταξιακών ε, συμφώνησαν όλοι ε, ότι δεν χωράνε βελτίωση και δεν χωράνε και εξυγχρονισμό μετά από γνωμοδοτήσεις των ε, εμπειρογνωμόνων και της Ευρατόμ έγιναν διάφορες δοκιμές και διάφορες ε, μελέτες και μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ γιατί είναι αντίστοιχοι οι αντιδραστήρες με τον μοιραίο αντιδραστήρα ε, του Τσερνόμπιλ και χαίρομαι ακόμα και σήμερα που ελήφθη τότε ομόφωνα αυτή η απόφαση να κλείσουν τα τρία εργοστάσια. Αλλά επίσης χαίρομαι και καλωσορίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να επομιστεί ένα μεγάλο τμήμα του κόστους ε, παροπλισμού και να συνεχιστεί αυτή η συμμετοχή γιατί επανειλημμένα έχει ληφθεί απόφαση για το ύψος της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποσόν και τώρα έχουμε μια πρόταση να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του παροπλισμού ε, του εργοστασίου Ιγναλίνα στη Λιθουανία. Ε, είμαι εγώ τώρα ε, η συγγήτρια για αυτό το θέμα και ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις, όσους ήρθαν και όσους δεν ήρθαν στην συνεδρίασή μας των σκιωδών. 53 είναι οι τροπολογίες, 18 δικές μου τη συζητήσαμε σε αυτή τη συνεδρίαση και σήμερα μπορώ να πω για τα σημαντικότερα θέματα που μας απασχόλησαν ότι η πλειονότητα των σκιωδών εισηγητών υποστηρίζει στην περίπτωση της Ιγναλίνα τη συγχρηματοδότηση και το ποσοστό να παραμείνει στο 86% και να μην μειωθεί. Επίσης μπορώ να πω ότι η πλειονότητα των σκιωδών εισηγητών επιθυμεί ρητά τα χρήματα αυτά που δίνονται στους Λιθουανούς να ε, αφιερωθούν αποκλειστικά στον παραπλησμό του εργοστασίου. Και επίσης πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η γνώση που έχουμε αποκομίσει που, που έχουν αποκομίσει από το παραπλησμό αυτό να ε, διαδοθεί για άλλες περιπτώσεις. Αλλά αν για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος οργανισμός, να βρεθεί νέα χρηματοδότηση. Γιατί στον προγραμματισμό για τον παροπλισμό δεν προβλέπεται αυτό. Όλα τα χρήματα που δίνουμε πηγαίνουν στον παροπλισμό. Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα με όλους τους εισηγητές, αλλά με την πλειοψηφία τους είναι ότι τα χρήματα αυτά που δίνουμε στους Λιθουανούς, στο επόμενο PDP, ε, ε, ε, συμφωνούμε οι περισσότεροι σκιώδεις και εγώ ότι το ποσό που προτείνουν οι Ιθουανοί, 780 εκατομμύρια, ε, είναι λογικό και αποδεδειγμένο ότι χρειάζεται με πολύ συγκεκριμένο και ακριβή σχεδιασμό. Ε, μετέβη και εγώ προσωπικά επιτόπου στην Ιγναλίνα και μίλησα ε, και με τους προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών και της κυβέρνησης και κανείς δεν αμφισβητεί αυτό το ποσό, τα 780 εκατομμύρια, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκδήλωσε εκεί ε, κάποιες ε, επιφυλάξεις ε, ως προς το λογιστικό σκέλος, το δημοσιονομικό δηλαδή, πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί το ποσό αυτό από το επόμενο PDP. Δεν αφισβητεί το ποσό. Στο μεταξύ ο συνάδελφος Λάγκεν, όπως άκουσα και από τις εξηγήσει του και διμερώς από συνομιλίες που είχαμε, έχει φέρει έναν άλλο ποσό, 683 εκατομμύρια, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Λάγκεν, αυτό βασίζεται στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις και υπολογισμούς για το κόστος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έχει πάρει τις αποστάσεις της από το ποσό αυτό, στο βαθμό που μπορώ εγώ να το παρακολουθήσω και να το αξιολογήσω και με έχει μπερδέψει λίγο η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την άλλη εβδομάδα θα συνεδριάσουμε και πάλι οι σκιώδεις συγητές και εγώ, αλλά νομίζω ότι το ποσό που δηλώνουν οι Λιθουανοί είναι περιστατωμένο, είναι τεκμηριωμένο, 780 εκατομμύρια. Είναι δύο οι αντιδραστήρες στη Λιθουανία που πρέπει να παραπληστούν, αλλά με χαρά να ακούσω την τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πιο πρόσφατη. Προσπάθησα να, σας, να, να βολιδοσκοπήσω τους δύο αρμόδιους επιτρόπους, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έχουν ακόμα συμφωνήσει με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ένα τελευταίο, το είπα και στην προηγούμενη έκθεση για τον Μποχουνίτσε και τον Κοσλοντούι, συμφωνώ απολύτως με αυτό που πρότεινε ε, ε, συνάδελφος Πούνσετ στην τροπολογία της ότι έχει ένα έκτακτο χαρακτήρα αυτή η χρηματοδότηση ε, και συνδέεται με τις συμφωνίες ένταξης των κρατών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παροπλισμού αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η πυρηνική βιομηχανία και ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τον παροπλισμό και τη διαχείριση των αποβλήτων. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, καθόλου δεν ισχύει ακόμα στα περισσότερα κράτη-μέλη κάτι τέτοιο. Αλλά η συγκεκριμένη χρηματοδότηση για την οποία συζητούμε είναι έκτακτη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει κανονικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Langen. Ο κύριος Λάγγεν, Ευχαριστώ πολύ. Ε, αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση για την οποία έχω διαφορετική γνώμη, γνώμη σε σχέση με την προηγούμενη. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά εργοστάσια με δύο τεράστια ε, μπλοκ. Έχει διαφορές λοιπόν από τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα έξοδα παροπλισμού με τις εκμείς του ελεκτικού ε, συνεδρίου θα ανέλθουν σε 5 δισεκατομμύρια 986 εκατομμύρια ευρώ στην Βουλγαρία 2 δισεκατομμύρια 697 εκατομμύρια και στη Βουλγαρία 2 εκατομμύρια 705 εκατομμύρια εδώ λοιπόν ε, το θέμα είναι η τάξη μεγέθους. Αυτό ε, πρώτον. Δεύτερον, η κυρία Χάρμς κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να ε, βρούμε ένα συμβιβασμό. Γι' αυτό οι προσπάθειές της με βρίσκουν θετικά προσκύμενα. Όμως ο εισηγητής έκανε προτάσεις οι οποίες δεν θα βρουν τη σύμφωνη γνώμη όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Έχουμε 8 πολιτικές ομάδες, 8 σκιώδεις εισηγητές, 8 άτομα δηλαδή. Αλλά δύο από τις ε, ομάδες αυτές είναι αρκετά μεγάλες ώστε αν ε, ενώσουν τις απόψεις τους να έχουν πλειοψηφία. Η βιομηχανία θέλουμε να έχει την ευθύνη. Κύριε Χάνης, δεν διαφωνώ μαζί σας. Στην περίπτωση της Ικναλίνα έχουν γίνει επισκευές 300 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Το 2008 πήγα και ο ίδιος ε, εκεί και συνάντησα τον αρχιμηχανικό ο οποίος μου είπε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και παρά τις επισκευές που έχουν γίνει πρέπει να παροπληστεί το εργοστάσιο οπωσδήποτε. Υπάρχει σίγουρα υποχρέωση που προκύπτει από τις ε, συνθήκες προσχώρησης. Όμως, λόγω του μεγέθους του εργοστασίου στην Ιγναλίνα πρέπει ε, να το θεωρήσουμε ε, εξαίρεση. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, η ευθύνη παροπλισμού ε, της Λιθουανίας ε, θα ανέλθει στο 14%, 14 ε, του κόστους και το 86% θα το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύμφωνα όμως με την άποψή μου και την άποψη του ΕΛΚ θα, μπορέσουν, ε, θα έπρεπε να ξεπεράσουμε αυτό το ποσοστό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, χρηματοδοτήσει ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό. Μπορούμε τώρα να δούμε τις λεπτομέρειες ε, και σε σχέση με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προτείνονται 525 εκατομμύρια ευρώ. Η κυρία Χάρμς προτείνει 80, 780 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει όμως να αναλογιστούμε τις διαστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν και το ποσοστό αυτό είναι τόσο υψηλό. Θα ήθελα όμως να, πω, ε, να ρωτήσω μάλλον την Επιτροπή εάν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία, νεότερες ε, πληροφορίες, να δούμε αν συμφωνούν αυτά τα ποσά. Σίγουρα υπάρχουν αποκλήσεις και αυτό το θεωρώ φυσιολογικό. Γι' αυτό λοιπόν, αν καταφέρουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση, δηλαδή ένα ποσό λίγο πάνω από αυτό που πρότεινε η κυρία Χάρμς. ...680 δηλαδή εκατομμύρια ευρώ προτείνω, μπορεί να είναι και 690, δεν πειράζει. Και, να, ε, και το ποσοστό χρηματοδότησης της κυβέρνησης της Λιθουανίας να είναι το πολύ 14%. Εάν μείνουμε σε αυτή την πρόταση, θα συμφωνήσουμε με απόλυτα με την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης της Λιθουανίας. Ο κύριος Κουρουμπάτσεφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι υπέρ της ε, αύξηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα παροπλισμού για τα πυρηνικά εργοστάσια. Χαίρομαι που ο κ. Λάγκερ έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την προηγούμενη και ότι θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να είναι το πολύ 40% μιλώντας για τη συμμετοχή της ε, Λιθουανίας, θα πρέπει να είναι 14% από την πλευρά της Λιθουανίας και 86% από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η περίπτωση της Ιγναηλίνα είναι εντελώ διαφορετική σε σχέση με αυτή της ε, Βουλγαρίας και της Σλοβακίας. Είναι αντιδραστήρις τύπου Τσερνομπίλ στην τη ε, Λιθουανία έχουν την, ομάδα, την μονάδα RBMK, ενώ στο Κοζοντού και στην Ποχούνιτσα έχουν ε, την μονάδα τύπου ΒΕΡ, που δεν είναι οι ίδιες ε, με τη συμμετεργοστάσια τύπου Τσερνομπίλ. Είμαι μηχανολόγος στο επάγγελμα και το γνωρίζω αυτό. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω την άποψη του να έχουμε συγκεκριμένα κονδύλια για την διάδοση πληροφοριών και γνώσεων που θα είναι ξεχωριστές από τη χρηματοδότηση για, για τον παροπλισμό. Υποστηρίζω την πρόταση του κυρίου Λάγκεν να αυξηθεί η χρηματοδότηση Ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να υποστηρίξει την πρότασή μας για αύξηση της χρηματοδότησης της 780 εκατομμύρια. Οι δύο αυτοί αντιδραστήρες την Ιγναλίνα θα πρέπει να κλείσουν το 2038, δηλαδή έχουμε 20 χρόνια μπροστά μας. Αν αναβάλουμε τη χρηματοδότηση Αυτό θα γίνει ακόμα πιο ακριβό με το πέρασμα του χρόνου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Πούνσετ. Από την άλλη, εμεί υποστηρίζουμε την αύξηση της χρηματοδότησης για το παροπλισμό της Ιγναλίνας στο 86% λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική δέσμευση της Λιθουανίας να ε, βάλει το υπόλοιπο 14%. Αλλά όπως και ε, άλλες πολιτικές ομάδες βάζουμε και όρους εμείς. Τα ποσά εκεί θα πρέπει να πηγαίνουν 100% για τον παροπλισμό. Αυτό είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος. Αυτό δεν αποκλείει ή δεν εμποδίζει να αναγνωρίσουμε και συμπληρωματικό ε, στόχο τη διάδοση των γνώσεων και των εμπειριών γιατί είναι πραγματικά ειδική φύσεω ο συγκεκριμένο παροπλισμό και μπορεί να βοηθήσει να κλείσουν και άλλα εργοστάσια σε κράτη-μέλη και ε, ε, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το 14% που δίνει η Λιθουανία. Το κόστος για το κλείσιμο και το παροπλισμό των πυρηνικών ε, εργοστασίων που γράφεται για ιστορικούς λόγους στη Συμφωνία Προσχώρησης του 2003 είναι ανδιαφυσβήτητο. Δεν το αμφισβητούμε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι μας αποκλείει από το να σκεφτούμε τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το κόστος που απορρέει. Κλείνουν τα εργοστάσια που είναι από τα παλαιότερα στον κόσμο. 75% των πυρηνικών εργοστασίων είναι ηλικία άνω των 30 ετών και πάνω από 90 εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κλείσει και μένουν χωρίς να παροπλιστούν εκεί. Έχουμε συμβαστικές τροπολογίες με τις οποίες συμφωνούμε και ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την αφοσίωσή της αλλά και τη γνώση της που θα βοηθήσει πολύ στην ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κόλλη Κόχιτς. ο κύριος. Κύριε Λάγκεν. Θα ομολογώ ότι με εκπλήξατε λίγο. Θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε σε αυτό το 14% που πρέπει να πληρώσει η Λιθουανία. Πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός θα είναι 0% το όλο ε, εγχείρημα θα γίνει σε 20 χρόνια. Ναι, εντάξει, τότε θα πρέπει να μιλάμε για μια συμμετοχή της λιθωνίας κατά 14%. Τώρα ας δούμε τι ακριβώς είναι ο παροπλισμός δεν μιλάμε μόνο για αντιδραστήρες, μιλάμε και για τα πυρηνικά κάψιμα. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν και τα πυρηνικά κάψιμα. Τι θα κάνουμε, θα τα διαθέσουμε, θα τα απορρίψουμε, εδώ θα υπάρχει συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Πρέπει να πω ότι με εκπλήξατε και με εκπλήξατε ευχάριστα κύριε Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Πάτσιτης. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ισχυώδεις εισηγητές και ο εισηγητής γνωρίζουν καλά το θέμα. 14 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε έχουν ληφθεί πολιτικές αποφάσεις και κάποιος είπε σήμερα έχετε υπογράψει μία συμφωνία. Βεβαίως δεν το συζητάμε αυτό. Αν δεν το είχαμε υπογράψει δεν θα είχαμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία πλευρά έπρεπε να το υπογράψουμε, από την άλλη είμαστε ευγνώμονες ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικά δεν μπορεί κανείς εύκολα να εξηγήσει τις αποφάσεις. Σήμερα όμως μιλάμε για θέματα ασφάλειας και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στη Λιθουανία, στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο πραγματικά ήταν πολύ επικίνδυνο. Σε ό,τι αφορά το παροπλισμό αυτών των πυρηνικών εργοστασίων, πιστεύω ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα ποσά για τον παροπλισμό. Γι' αυτό με εξέπληξε η πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση. Μιλώντας για την Ιγναλίνα και αναφερόμενη στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ήταν δύσκολο να πείσουμε την Επιτροπή πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το πυρηνικό αυτό εργοστάσιο. Σιγά σιγά όμως Είχαμε περισσότερες γνώσει. τα μέλη τη Επιτροπής Προπολογισμού πήγα στη Λιθουανία, είδα πώ ακριβώ έχουν τα πράγματα και βλέπουμε ακριβώ τι συμβαίνει. Θα πρέπει να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αυτό απαιτείται για την ασφάλεια όχι μόνο στη Λιθουανία αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποθήκευση των καυσίμων γίνεται εκεί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν αποθηκευτικοί χώροι. Γιατί είναι πιθανόν να υπάρξει μόλυνση των Λιθουανών και των, και των όμορων χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που καταλάβετε ότι τα πυρηνικά εργοστάσια είναι επικίνδυνα, ότι τα ραδιενεργά απόβλητα, είναι επικίνδυνα και για το λόγο αυτό χρειάζεται απερκής χρηματοδότηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή καταρχάς. Η στάση της ήταν λίγο εχθρική. Αργότερα οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έμαθαν πολλά, πήραν μέρος στην όλη διαδικασία και τώρα νομίζω ότι αυτός ο γενικός συμβιβασμός που καταλήγει στο ποσοστό χρηματοδότησης 14% είναι αποδεκτό και δεν θα αφιστούμε προσπαθειών προκειμένου να εφαρμοστεί το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για τη Λιθουανία και για τις όμονες χώρες προκειμένου να νιώθουν ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάσιμο Γκαρίμπα από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ε, ευχαριστώντας τον εισηγητή Θυμάμαι ότι αυτή η κατάσταση, αυτό το διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, ε, έκλεισε, ήταν προπόθεση να κλείσει και η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Φέτος ε, υπήρξε μια παρέμβαση στους δύο αντιδραστήρες και τα καύσιμα αποθηκεύονται σε αποθηκευτικούς χώρους. Η πρόκληση για το επόμενο πλαίσιο, είναι η πλήρης, ο πλήρης ε, ε, παροπλισμός σε μία τρίτη δράση αυτής της κλίμακας. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι η Ένωση συνέβαλε οικονομικά από το τέλος αυτής της οικονομικές περιθώρους καταβάλλοντας 1,9 δις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σημεία που εστέθησαν από τον εισηγητή, πραγματικά υπάρχει ένα κενό οικονομικό και το οποίο αναγνωρίζει και η Επιτροπή και οι αρχές Λιθουανίας για την περίοδο 2020 μέχρι 2028 που επεκτείνεται πολύ περισσότερο και αφορά 1,3 δις. Αυτός ο υπολογισμός είναι λογικός και για την Επιτροπή και για την κυβέρνηση της Λιθουανίας. Υπάρχει επίσης ως μέρος του τρέχοντος κανονισμού ένα πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε και συμφωνήθηκε το 2014 και για την επόμενη ε, περίοδο προβλέπει χρηματοδότηση 502 εκατομμυρίων. Αυτό αντιστοιχεί στο ποσό που προτάθηκε από την Επιτροπή. Επιτρέψτε μου επίσης ε, να σας θυμίσω ότι το ποσό αυτό βασίζεται στην δυνατότητα της Λιθουανίας να απορροφήσει αυτή τη χρηματοδότηση για ε, παροπλισμό. Βεβαίως μετά από αυτή την οικονομική περίοδο παραμένει ένα κενό και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των αξιότιμων μελών στο ότι για πρώτη φορά στην τον προτινόμενο κανονισμό υπάρχει αναγνώριση της δομής αυτού του προγράμματος και του γεγονότος ότι η Επιτροπή αναμένει ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί και μετά το πέρας του τρέχοντος ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αρκετά μέλη αναφέρθηκαν στο θέμα των γνώσεων, των κοινών γνώσεων. Όταν κοιτάξετε την άλλη πρόταση, την πρόταση για την οποία είναι εισηγητής ο κύριος Κουρούμπατσεφ, θα δείτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που προτείνεται για παροπλισμό και υπάρχουν και τα χρήματα που αφορούν τη διάδοση γνώσεων. Η Επιτροπή, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση θα μπορούσε να υποβληθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο σημείο του οποίου υπάρχει συμφωνία αφορά την συγχρηματοδότηση 14% η οποία υποστηρίζεται από πολιτικές δηλώσεις στη Λιθουανία. Επιτρέψτε μου να τονίσω ένα σημείο. Υπάρχει ένα ανώτατο σημείο για το πρόγραμμα και αυτό όμως δεν αποκλείει το να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν πλήρως ορισμένες δράσεις κατά 100% όπως εξάλλου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάγκεν. Μία σύντομη ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε δύο προτάσει σα αυτή τη στιγμή. Είναι ρεαλιστικέ ή δεν έχει κανένα νόημα να τι συζητάμε. Μετά από αυτό που είπατε, <laughs> δεν ξέρω τίποτα πια. Έχει νόημα δηλαδή να αυξήσουμε τη συγχρηματοδότηση ή όχι. Τι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι η λύση. Ε, να το πω κι αλλιώ. Αν θέλω να, κοροϊδέψω, να με κοροϊδέψει κάποιο, μπορώ να κοροϊδέψω κι εγώ τον εαυτό μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση τον Ιούνιο για τα τρία αυτά προγράμματα και είναι μια πρόταση η οποία, όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω, βασίζεται στα τρέχοντα ποσά συγχρηματοδότησης. Το ερώτημα που προέκυψε στο στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν νομίζω πως ε, αφορά τις άλλες δύο, είναι τι ποσό θα διατεθεί σε αυτό το πολιτές χρηματοδοτικό πλαίσιο και τι θα μείνει για το επόμενο. Ή εάν θα χωριστεί το ποσό με διαφορετικό τρόπο. Η τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 552 εκατομμύρια ευρώ να υπενθυμίσω, λαμβάνει υπόψη τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο έχει σήμερα. Ωραία, τα τελικά σχόλια θα γίνουν φυσικά από την εισηγήτρια. Ε, εννοείται. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κρουμπάσεφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζεκ. Αναρωτιέμαι και θέλω να ξανακάνω την ερώτηση που έκανε ο κύριος Λάγκεν. πώς μπορείτε σε αυτή την περίπτωση να έχετε ένα ανώτατο όριο 80% αλλά κάποιες δραστηριότητες να τις χρηματοδοτήσετε κατά 100%. Όταν το ανώτατο όριο είναι το 80% πώς φτάνουμε στο 100%. Όταν το ελάχιστο είναι 80% τότε μπορείς να χρηματοδοτήσεις 100% κάτι. Τέλος. 552 εκατομμύρια θέλετε, 683 εκατομμύρια θέλετε ή 708. 80, 780. Ποιο από τα τρία ποσά ισχύει, ποιο από τα τρία είναι το καλύτερο. Η ε, κυρία Χάρμς έχει το λόγο. Από πού να αρχίσω. Λοιπόν, δεν είμαι τόσο εξοργισμένη όπως ο κύριος Λάγκεν, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι κάπως μπερδεύομαι καμιά φορά με όλα αυτά τα διαφορετικά νούμερα που ακούμε για το συγκεκριμένο σκέλος του παροπλισμού στην Ιγναλίνα, το οποίο συζητούμε τώρα. σχέδιο για το οποίο οι Λιθουανοί μας υπέβαλαν λεπτομερέστατη έκθεση. Είναι το πιο ακριβό κομμάτι αυτού του παροπλισμού, διότι και οι δύο αντιδραστήρε ε, πρέπει να παροπλιστούν. Επαναλαμβάνω, και οι δύο αντιδραστήρε. Οι υπολογισμοί που έχουν δοθεί από την ε, διοίκηση του εργοστασίου της Συγναλίνα στο μεταξύ έχουν χαρακτηριστεί αξιόπιστοι και αντικειμενικοί και χαρακτηρισμένοι από επαγγελματισμό από όλους τους διεθνείς φορείς. Δεν αμφισβητείται ε, τίποτα. Εάν αρχίζει και αμφισβητείται το ποσό των 780 εκατομμυρίων ευρώ, τότε αμφισβητείται και όλο το πρόγραμμα παροπλισμού της Ιγναλίνα. Εάν αμφισβητούμε δηλαδή τις ανάγκες παροπλισμού, τότε αμφισβητούμε και την ανάγκη παροπλισμού του δεύτερου αντιδραστήρα. Η άποψη που, που σχημάτισα Άποψη την οποία συμμερίζεται και ο κύριος Νόβακ από την ε, EBRT, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και για τον παροπλισμό στο Τσερνόμπιλ. Είναι πως τα νούμερα στέκουν. Είναι σωστά. Τώρα, να αρχίσουμε να ψάχνουμε και να ψυρίζουμε το καθετή και να ε, ε, επανεξετάζουμε το παραμικρό και να αμφισβητούμε δηλαδή τους ε, υπολογισμούς των Λιθουανών, τότε δεν νομίζω να δοθεί ποτέ πράσινο φως. Μου φαίνεται πως όλο το εγχείρημα θα γίνει πολύ ακριβότερο εάν αναβάλουμε τον παροπλισμό του δεύτερου αντιδραστήρα για το μέλλον τότε οι Λιθουανοί θα αποκτήσουν πρόβλημα. Για παράδειγμα, το προσωπικό που εργάζεται σήμερα στον αντιδραστήρα, το οποίο είναι καλά καταρτισμένο, θα μείνει άνεργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε ένα πιθανό πρόβλημα, τη δυνατότητα απορρόφησης ε, των Λιθουανών. Το κοιτάξαμε και η ικανότητα απορρόφησης ε, στη Λιθουανία τα τελευταία χρόνια απεδείχθη αρκετά υψηλή, 100 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και αυτό ακολουθώντας σχέδιο, το οποίο σχέδιο καταρτίστηκε και στηρίχθηκε από όλους. Ήταν ένα σχέδιο που ε, είχε υπολογίσει κόστος 100-130 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για, για όλη την διαδικασία του παροπλισμού του εργοστασίου. Κατά την προσωπική μου άποψη θα χρειαστούμε συνάντηση σκιωδών. Αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Όμως για μένα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρνηθούμε και να αμφισβητήσουμε αυτό το ποσό των 780 εκατομμύριων, ευρώ. Και νομίζω πως οφείλουμε να στηρίξουμε την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Κατανοώ ε, ότι είναι απαραίτητη η συνεδρία συνεδρίαση σκιωδών, όπως πάντα. Α, συγγνώμη, Πρόεδρε, ε, λέει η κυρία Χάρμς, αύριο, αύριο, όχι την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα, αύριο είναι η συνεδρία του σκιωδών εισηγητών. Ο κύριος Λάγκεν. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια πρόταση μετά τα λεγόμενα της κυρίας Χάρμς εσείς ως πρόεδρος της Επιτροπής Ήτρε, γιατί αποφασίζουμε στις 3 Δοδεκάτου, μπορείτε να στείλετε επίσημη επιστολή στους δύο αρμόδιους επιτρόπους, Ότιγκερ και Άρια Κανιέτε, για να μας ενημερώσουν ε, ποια, πού είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρόταση της Λιθουανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν υπάρχει δυνατότητα να εξευρεθεί μια λύση. Νομίζω αυτό θα ήταν μια λογική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως χρειάζεται να κάνει κάποια διορθωτικά σχόλια. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι εκπροσωπείται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Χάμς. Είχα πολύ έντονη συνομιλία με τον κύριο Έτιγκερ αμέσω μετά το θέρος και του είπα ε, τι είχα δει στην Ιγναλίνα, του ανέφερα τα πεπραγμένα της επίσκεψης και εκεί συμφωνήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτο θα πρέπει να είναι αξιόπιστη στα μάτια των Λιθουανών και να συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο για την Ιγναλίνα και τη Συμφωνία ε, Προσχώρησης, τη συνθήκη. Και δεύτερον, κατάλαβε και ο κύριος Σιώτιγκερ ότι δεν θα πρέπει να διακοπεί ούτε να καθυστερήσει ε, ο προγραμματισμός γιατί αυτό θα επιφέρει ένα επιπλέον κόστος. Και ξέρω ότι δύο επιτροποί συντάσσουν ε, επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ε, εισηγητές αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν συμφωνήσει για το περιεχόμενο της επιστολής. στο τέλος μάλλον θα είναι πολύ πολιτική η απόφαση, αλλά δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε αντικείμενο ε, της ε, διαπραγμάτευσης ή του παζαριού αυτού. Αλλά να πάρουμε την απόφαση βάσει των πληροφοριών που λαμβάνουμε και τον οικονομικό σχεδιασμό. Και όχι στα κουτούρου Μάλιστα, όπως βλέπετε κάναμε μια ευρεία και πολύ βαθιά συζήτηση στην Επιτροπή μας. Τα υπόλοιπα παρακαλώ να συζητηθούν στις συνεδρίες των σκιωδών, ως ήθιστε. Εκεί είναι ο κατάλληλος τόπος. 21 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, ενώ στην Ολομέλεια στη... το Γενάρη. Τελευταίο θέμα για σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Αναδιατύπωση. Our reporter. Ε, μας είναι ο κύριος Νεοκλής Σιλικιώτης. Και έχουμε 323 τροπολογίες. 58 του εισηγητού. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ Εσωτερικής Αγοράς ήδη ενέκρινε τη γνωμοδότησή τους με 93 τροπολογίες, ενώ οι δύο οι επιτροπές ΚΑΛΤ και ΛΥΜΠΕ θα ψηφίσουν στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Δηλαδή θα έχουμε και άλλες τροπολογίες από την ΚΑΛΤ και τη ΛΥΜΠΕ. Από την ΙΜΚΟ σας είπα 93. Με τις δικές μας, συν, 323. Το λόγο έχει ο κύριος Ηλικιώτης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές της έκθεσης καθώς και τους συνεργάτες τους και βεβαίως τα ε, προσώπους της γραμματείας της Ίντρα για την άψογη συνεργασία που έχουμε. Είμαι σίγουρος όπως ο στόχος είναι κοινό και με συλλογική δουλειά θα επιτύχουμε τη βελτίωση του κειμένου προσπερνώντας τι επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί βοηθούν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός συμβαστικού κειμένου που θα μας εκφράζει όλους, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, αλλά και θα καθησυχάζει και τις ανησυχίες μας. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε πως τα ανοιχτά δεδομένα θα αποφέρουν πραγματικό όφελο στους ανθρώπους και την κοινωνία και θα αξιοποιούνται κυρίως για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των νέων αναδυόμενων επιχειρήσεων. Και όχι μονάχα με, να αξιοποιούνται από τις μεγάλες πολυεθνικές όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Εξάλλου οι μεγάλες εταιρείε έχουν τα οικονομικά μέσα ε, να παίρνουν όλες τις προφορίες. Αυτός ακριβώς είναι και ο βασικός στόχος των συμβαστικών τροπολογιών που έχουμε ετοιμάσει μέχρι τώρα. Όσον αφορά τα δεδομένα υψηλής αξίας, προχωρήσαμε σε αυτό που είχαμε πει εξ αρχής, στην κατάθεση συγκεκριμένη λίστα με κατηγορίε συνόλων δεδομένων υψηλή αξία. Στην πρόταση μα προβλέπεται πω η Κομισιό θα μπορεί να προσθέσει και νέε κατηγορίε εφόσον προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψει όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τα δεδομένα υψηλή αξία έχουν παραχθεί με δημόσιο χρήμα και πρέπει να οθεί στην κοινωνία. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δημοσιοποιηθούν δεδομένα που θα φέρουν σε δυσμενή θέση είτε των δημόσιων τομέα, είτε τους κρατικούς, τους δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι παλεύουν και τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες παλεύουν σε δύσκολες συνθήκε έχουν να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά. Γενικότερα, διότι όσον αφορά τι δημόσιε επιχειρήσει και τη συμπερίληψή του στο πεδίο εφαρμογή τη λόγω οδηγία, σε μια προσπάθεια συμβιβασμού και συγκερασμού των διαφόρων απόψεων που ακούστηκαν, οφείλουμε να συμπεριλάβω στο κείμενο τέτοιε πρόνοιε που να διορθώνουν τι σεβαρέ τροβλώσει οι οποίε δημιουργούνται, κατά την άποψή μα, με το κείμενο που προτείνει η Κομισιόν. Εφόσον όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού, θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να βελτιώσουμε το κείμενο για να μην ενταθούν ακόμα περισσότερο οι άνισοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις περιπτώσει, όπου <clears throat> λειτουργούν και ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά. Ε, Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ακόμη μια φορά την ανάγκη να στηρίξουμε οικονομικά ω Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τεχνικά, δημόσιε επιχειρήσει, ιδιαίτερα σε αυτέ που βρίσκονται ε, σε μικρούς δήμους οι οποίοι θα καλεστούν να υλοποιήσουν αυτή την οδηγία ώστε να έχουμε ε, πραγματικά το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι απόν. Είναι ο κύριος Μπόνη. Και με παρακάλεσε να διαβάσω την άποψή του. Λοιπόν, αρχίζω την ανάγνωση. Η οδηγία PSI είναι ένα βήμα για τη νέα χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και αυξάνει όλο και περισσότερο στη σημασία της γιατί είναι πηγή για καινοτόμες υπηρεσίες όσο και προϊόντα. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι ο κανονισμός αυτός έχει στόχο να διευκολύνει την εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με εναρμόνιση ε, των βασικών προϋποθέσεων έτσι ώστε ε, οι πληροφορίε του δημοσίου τομέα να είναι προσβάσιμες σε χρήση και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξή τέσσερα. Ε, νέα προϊόντα και υπηρεσίε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθάρρυνση της διεθνώριακή χρήση των πληροφοριών αυτών ε, και δεδομένων, πρόληψη της στρέβλωσης του ανταγωνισμού για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και με μηχανισμό αποζημίωση όταν αυτό χρειάζεται. Και το τέταρτο σημείο και τελευταίο είναι περιορισμός των εξαιρέσεων που επιτρέπουν σε οργανισμούς ε, του δημοσίου τομέα να επιβάλλουν χρέωση για να καλύψουν κάποιο περιφερειακό κόστος. Προσβλέπει στη συνεργασία με τους σκιώδες εισηγητές ο κ. Μπόνη και προτείνει πρόσβαση και εκ νέου χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα με την πολιτική Open Data της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο για τη διαφάνεια του δημοσίου τομέα και τη χρήση ε, υποστηρικτικής τεχνολογίας από τους φορείς του δημοσίου. Ταυτόχρονα αυτό βοηθάει και τις δημόσιες και τις ε, ιδιωτικές υπηρεσίες και τη γνώση των πολιτών για να παίρνουν αποφάσεις ε, καλύτερα ενημερωμένοι. Και για μελλοντική συνεργασία ένα δεύτερο σημείο επίσης που προτείνει ο κύριος Μπόνη είναι τα δεδομένα υψηλής αξίας να ε, ανοίξουν στην πρόσβαση ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την αναδιατύπωση, ιδιαίτερη σημασία να υπάρξει ένας κατάλογος κατηγοριών δεδομένων υψηλής αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να έχουμε ε, μια εναρμόνιση και μια συνεκτική προσέγγιση. Ο κατάλογος αυτός δεν θα πρέπει να είναι εξαντλητικός και μπορεί να συμπληρωθεί ή να συμπληρώνεται κάθε φορά με κατεξουδότηση πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσθέτει νέες κατηγορίες όταν χρειάζεται αυτό. Αυτά λέει ο κύριος Μπόνι. Και τώρα προχωρούμε στον επόμενο σκιώδη συγητή που είναι ο κύριος Πέντερσεν από τους Φιλοελευθέρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος εγώ, διότι πιστεύω ότι συμφωνούμε και όλοι οι σκιώδες, τουλάχιστον για τις γενικές προθέσεις και τη φιλοδοξία αυτής της σημαντικής πρότασης για την εκ νέου χρήση προφοριών του δημοσίου τομέα. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό στην ανάπτυξη των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, η γενική φιλοδοξία και η γενική πρόθεση αυτής της σημαντικής πρότασης με βρίσκει όλους ε, σύμφωνους. Από πλευράς μας ε, προσβλέπουμε πάρα πολύ στην πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών ε, εισηγητών αύριο Μπορεί να χρειαστεί να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες και μπορεί να χρειαστεί και να διαφωνήσουμε, γιατί όχι στην ψηφοφορία σε συγκεκριμένες ε, τροπολογίες. Γενικώ όμως πιστεύω ότι συμφωνούμε ως προς την κατεύθυνση και τη φιλοδοξία, επαναλαμβάνω. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε, άμα θέλετε, και τη συμπερίληψη ιδιωτικών φορέων όταν παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Γενικώ συμφωνούμε για τις προθέσεις, για τη φιλοδοξία. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση και με χαρά ε, θα έχουμε αύριο την πρώτη συνεδρία στις Σκηδών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ρέντα από πλευρά των Πρεσίν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρώτη ομάδα συμβιβαστικών τροπολογιών και προσβλέπω επίσης την αυριανή συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών. Είναι φιλόδοξη η ατζέντα μας και πρέπει να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την σημαντική νομοθεσία πριν λήξει η θητεία μας. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση για τη διαδικασία. Όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια νομοθεσία είναι πολλές φορές δύσκολο όταν υπάρχουν πολλές συμβαστικέ προτάσεις για το ίδιο άρθρο. Προτείνω λοιπόν να έχουμε τέσσερις ή πέντε συμβαστικέ τροπολογίες για το, για το κάθε άρθρο. Στην Επιτροπή που ήμουν η ε, εισηγήτρια είχαμε πολύ καλή εμπειρία στην ΕΜΚΟ λοιπόν ε, για, με αυτήν την ε, μέθοδο. Πολλές φορές είναι σημαντικό να μην αλλάζει η πρόταση της ε, Επιτροπής. Σε αυτό δηλαδή συνίσταται ο συμβιβασμός. Το συνολικό αποτέλεσμα πιστεύω θα είναι πιο συνεκτικό μετά την ψηφοφορία και έτσι θα μπορέσουμε όταν εισέλθουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να ζητήσουμε αυτά που θέλουμε. Αυτή τη στιγμή βλέπω να λείπει συνοχή σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, στις ε, δημόσιες ε, επιχειρήσεις να πω καταρχά ότι είδαμε με μεγάλη μα χαρά ότι ο συγητή συμπεριέλαβε τι δημόσιε επιχειρήσει στην συμβαστική τροπολογία 1 και τι ιδιωτικέ επιχειρήσει, εφόσον αυτέ ε, πληρούν συγκεκριμένε προποθέσει. Όμω στη συμβαστική 2 και 3, οι οποίε αφορούν το ίδιο άρθρο, γίνονται εξαιρέσει για δημόσιε επιχειρήσει. Αυτέ οι εξαιρέσει είναι τόσο γενικέ που νομίζω πω δεν θα ε, μείνει τίποτα στην ουσία στο τέλος όλα τα έγγραφα των επιχειρήσεων ίδρυυσης ηλεκτρισμού, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών ή μεταφορών θα εξαιρούνται και αναρωτιέμαι λοιπόν τι θα μείνει όταν ε, αναφερόμαστε στις, ε, στα δεδομένα των δημόσιων επιχειρήσεων. Όταν επίσης εξαιρούνται ολόκληροι τομείς για λόγους ασφαλείας, που νομίζω πως ήταν ο αρχικός σκοπός της Επιτροπής, ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, να καταλήξουμε δηλαδή σε μια περίπτωση όπου όταν μια εταιρεία ηλεκτρισμού έχει έγγραφα τα οποία είναι βέστητα από πλευράς ασφαλείας και δεν πρέπει να διατεθούν στο κοινό, τότε όλος αυτός ο τομέας θα εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Νομίζω πως δεν είναι αυτή η πρόθεση της Επιτροπής, γι' αυτό οι συμβαστικές προτάσεις 2 και 3 για μένα χρειάζονται λίγο παραπάνω ε, δουλειά. Επίσης, ε, χαιρόμαστε πολύ για το ότι ο εισηγητής έχει συμπεριλάβει το παράρτημα των ε, ομάδων δεδομένων υψηλής αξίας και προτίθεται να τροποποιήσει το παράρτημα. Θεωρούμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει όχι μόνο τις κατηγορίες αυτών των ομάδων δεδομένων, αλλά και τις συγκεκριμένες ομάδες που θα χαρακτηρίζονται ως ομάδες υψηλής αξίας. Διαφορετικά τα κράτη-μέλη δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι πρέπει να συμπεριληφθεί και τι όχι. Τώρα, αυτά τα δεδομένα υψηλή αξία, ε, ω προ αυτά, νομίζουμε πω η πρόταση είναι αρκετά καλή, ο κατάλογο είναι καλό, θα θέλαμε όμω να προσθεθούν και κάποιε εθνικέ λίστε με την νομοθεσία, διότι δεν δημοσιεύουν δωρεάν όλα τα κράτη-μέλη την νομοθεσία του και θεωρούμε ότι κάθε πολίτη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει του νόμου του κράτου του. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα με τις ομάδες δεδομένων υψηλής αξίας. Τώρα, όσον αφορά τα APIs, καλωσορίζουμε την ε, αναφορά στον πραγματικό χρόνο real time, χωρίς καθυστερήσεις στην προσβασιμότητα των δεδομένων αυτών. Επίσης, οι τροπολογίες για την οδηγία βάσεων δεδομένων ε, που έχουμε υποβάλει θα θέλαμε να ληφθούν υπόψη διότι νομίζουμε πως είναι αρκετά σημαντικές. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ πρέπει να ενισχυθεί. Προσβλέπουμε λοιπόν και εμείς τις συζητήσει πάνω συμβαστικέ τροπολογίε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμβιβαστούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία της πρότασης, διότι έτσι θα καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό κείμενο που θα μας δώσει μια ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταμποράνο για το EFTD. Κυρία Πρόεδρε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτοί που προέρχονται από τον ιδιωτικό δημόσιο τομέα να χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή που θα μπορούσαν να συμβάνουν όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό και απασχόλησης αλλά και σε επίπεδο περιβαλλοντικό. Προκειμένου να μπορέσει να γίνει αυτό είμαστε σαφείς σαφώς υπέρ μιας συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών χωρίς να υπάρχουν πολλές εξαιρεσει. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διαφυλακτεί αυτό ως κοινό αγαθό και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ξεπεραστεί η ε, ψηφιακή κυριαρχία του δημοσίου. Το δημόσιο θα πρέπει να ξεπεράσει την αντίστασή του στην πρόσβαση των δεδομένων. Το δημόσιο θα πρέπει να μπορεί να στηριχτεί σε μια συγκεκριμένη υποστήριξη που επιτρέπει την κατάρτιση και την ε, ε, ύπαρξη δεδομένων. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε στο δημόσιο τη δυνατότητα πρόσβαση και κρίση δεδομένων που παράγονται από τι επιχειρήσει, δημόσιε επιχειρήσει. Και αυτό ανεξάρτητα από τη δημόσια ιδιωτική φύση μια επιχείρηση. Ε. δεν είμαστε μόνο υπέρ τη ε, διατήρησης του πεδίου εφαρμογής, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ε, αλλά είμαστε υπέρ του να συμπεριληφθούν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όταν παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο. Αυτό συμφωνεί με αυτό που προκύπτει από το Digital Transfiction Plan που ε, αφορά την, το αστικό χρονοδιάγραμμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είμαστε πεπισμένοι ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η χρήση των δεδομένων των ερευνών σε συγκεκριμένους τομείς που χρηματοδοτούν Τούντε εν μέρη ή καθ' ολοκληρία από δημόσια κονδύλια. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση Connect. Ο κύριος Ιβο Βόλμαν. Yes, thank you, Chair. And I would like to... Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και, για, και τα μέλη για τη συζήτηση και για τις τροπολογίες. Εδώ φαίνεται η σημασία που έχουν για την οικονομία, ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνία, αλλά και είναι και μια πηγή καινοτομία. Θα ήθελα να τονίσω μερικά σημεία. Πρώτον, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τη γενική κατεύθυνση της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα για τις ομάδες δεδομένων υψηλής αξίας. Κατανοώ ε, την επιθυμία να υπάρξει ένα πλαίσιο για τον κατάλογο σε κατηγορίες και όσο παραμένει ανοιχτός ο κατάλογος δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την πρόταση αυτή. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Άλλος τομέας είναι η σημασία του να έχουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ε, για διάφορες διαδραστικές έτσι, επιφάνεις, interfaces, διεπαφές και θα αναπεριοριστούν οι ε, εξαιρέσεις ε, για την κάλυψη μόνο του περιθωριακού κόστους. Για τις δημόσιες επιχειρήσεις σημειώνουμε πόσες ε, είναι οι τροπολογίες και σε ό,τι αφορά τις ΔΕΚΟ, τους οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας, είναι πραγματικά κρίσιμη τομής για την οικονομία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ένα σενάριο που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των δημοσίων επιχειρήσεων και την ανάγκη να υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού. Ε, κάτι άλλο τώρα για την ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια και τους, ε, τις βασικές ε, υποδομές της δημόσιας. Τα είπε η κυρία Ρέντα, βεβαίως θα πρέπει να προστατεύονται, αλλά θα πρέπει να βρούμε και την κατάλληλη διατύπωση για να μην καούν και τα χλωρά μαζί με τα ξερά γιατί υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξαιρούνται όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσει που δεν έχει νόημα ή δεν είναι στι προθέσει μα. Κάποιε από τι τροπολογίε ασχολούνται με κάποια στοιχεία τη οδηγία που δεν είναι ε, τμήμα τη αναδιατύπωση και υπάρχει κίνδυνο οπισθοδρόμηση σε κάποια στοιχεία σε σχέση με τα όσα ήδη έχουν συμφωνηθεί το 2013. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η οδηγία σταδιακά έχει εξελιχθεί και διαδοχικά έχουμε νέες ε, εκδοχές. Βεβαίως θέλουμε οι συζητήσεις σας να ε, οδηγήσουν σε ένα επίπεδο φιλοδοξίας αντίστοιχο με της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ακούσαμε προηγουμένως. Ελπίζω οι συνομοθέτες να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία, την οποία θα πλαισιώνουμε και θα παρακολουθούμε κι εμείς. Δεν ξέρω, ο κύριος Ηλικιώτης, αν θέλει να πάρει το λόγο και πάλι, παρακαλώ για τα τελικά καταληκτικά σχόλια. Πρώτα θα είμαι και εγώ πολύ σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω του ε, σκιωδησηγητέ για τι απόψει του ε, και να πω ότι βεβαίω υπάρχουν ζητήματα που έχουμε διαφορετικέ προσεγγίσει, όπω και με την Επιτροπή. Να πω ότι ε, ίσως το ε, πιο κέριο ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι ο τρόπος που θα μεταχειριστούμε τις δημόσιες επιχειρήσεις. Είπα και στην αρχική παρέμβαση θα πρέπει να διαμορφώσουμε ίσους κανόνες και δίκαιους κανόνες σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Ε, επειδή είχα την ευκαιρία να έχω επαφή με πάρα πολλούς ε, οργανισμούς από πολλές χώρες ε, και ομίλους ιδιαίτερα διαδημοτικές ε, οργανώσεις που λειτουργούν δημόσιες επιχειρήσεις, δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να ανταγωνισμό. Εάν υπάρχει λογική και θέλω να πω σε ό,τι αφορά του προτάσει συμβαδίου, επειδή αναφέρθηκε η συνάδελφο Ρέτα, για τη συμβασμό 1 και 2 και 3, να πω ότι εάν δεν συμπεριληφθούν ιδιωτικέ επιχειρήσει, τότε θα πρέπει να υπάρξουν μεγάλε εξαιρέσει. Ε, δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα φέρουμε του δημόσιου οργανισμού σε μειονεκτική θέση σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Άρα είναι δύο ζητήματα που πρέπει να τα δούμε μαζί ή συμπεριλαμβάνουμε και τι ιδιωτικέ επιχειρήσει και διαμορφώνουμε ίσου καλού ανταγωνισμού, ή ε, οδηγούμαστε να εξαιρέσουμε ε, ειδικότερα στοιχεία εκείνα που είναι εμπορεύσιμα, που μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν οι ανταγωνιστέ σε βάρο των δημόσιων επιχειρήσεων. Ε, τα λέω έτσι γιατί ε, τα πράγματα είναι κατά την άποψή μου πολύ ξεκαθαρά. δεν θα μπω σε περισσότερο λεπτομέρειε ό,τι αφορά το παράρτημα ε, για τις ε, κατάργων υψηλή αξίας. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ως συνομοθέτης ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει εισήγηση, γι' αυτόν κάνει και την εισήγηση. Βεβαίως θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή σε ένα ανοιχτό κατάλογο να μπορεί να συμπληρώνει αυτόν τον κατάλογο με κατεξουδότηση πράξη και εδώ πρέπει να είναι και η δική μας η προσπάθεια. Πιστεύω ότι ναι, ε, το βασικό κατεύθυνση τη ε, οδηγία αυτή πρέπει να υλοποιηθεί για να δώσουμε τη δυνατότητα σε μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, σε επιχειρήσει, αναδυόμενε επιχειρήσει, startups, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που θα βοηθήσουν αυτά τα δεδομένα να αναπτυχθούν και να δώσουν όθηση και στη δράση, τη δραστηριότητα του αλλά και στην ίδια την οικονομία και την κοινωνία. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη πάντοτε ότι ε, ευθύνη μας ως Ευρωκοινοβούλιο είναι να παρεμβαίνουμε ώστε να δημιουργούνται δίκαιοι κανόνες για όλους. Ε, και θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αύριο ε, θα έχουμε συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά ώστε στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει στις 3 του Δεκέμβρη δηλαδή να έχουμε την έκθεση ενώπιον της Επιτροπής για να ψηφιστεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Θαυμάσια. 3 Δεκέμβρη ψηφίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας, στην Ολομέλεια, πάλι το Δεκέμβριο, μάλλον, στο Στρασβούργο, μέσα Δεκεμβρίου, διάφορα. Συνάδελφοι, έχουμε προσεχή συνεδριάσεις. 21 Δεκάτου το πρωί και το απόγευμα και το αυτό για τις 22 Δεκεμβρίου, πρωί και απόγευμα. 14 ώρες και μισή θα είμαστε μαζί. Τεράστια συνεδρίαση, ευχαριστώ. Ε, καλή συνέχεια για τις επόμενες ημέρες.